So, dear colleagues, I think it's... Uh, Αγαπητοί συναδελφοί, είναι 3 και 4. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν. Το πρώτο θέμα που συζητούμε σήμερα το απόγευμα είναι το σημείο 9 της ημέρησης διάταξης για την εμπορική πολιτική και την άγρια πανίδα, η συγητής μας για το θέμα αυτό, είναι η κυρία Μακλάρκιν, η οποία είναι παρούσα εδώ φυσικά, και το θέμα μας είναι η ευρωπαϊκή πολιτική ενώπιον της ανάγκης προστασίας της αγρίας πανίδος. Και έχουμε πολλούς ε, διακεκριμένους καλεσμένους. Δύο πάνελ έχουμε. Πρώτον για τη δημιουργία του πλαισίου πολιτικής για το εμπόριο και την, τις αρχέ και το δεύτερο για να δούμε περισσότερο σε λεπτομέρεια τις ε, προκλήσεις που συναπτώνται με την προστασία της άγριας ζωής και για την ε, δίωξη της λαθεμπορίας αγρίας πανίδος. Καλώς ήρθατε λοιπόν διακεκριμένοι καλεσμένοι και πρωτού ξεκινήσουμε, ξεκινήσουμε με το πρώτο πάνελ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μακλάρκιν, την εισηγήτριά μας το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω κι εγώ καλωσορίζοντας τους φιλοξενούμενους που είναι εδώ σήμερα Κάποιοι από αυτούς έκαναν τεράστιες, διένυσαν τεράστιες αποστάσεις για να πάρουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση, την τόσο σημαντική. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που βρήκατε το χρόνο να έρθετε εδώ, το εκτιμούμε δεόντως. Ίσως κάποιοι να εκπλήσεστε, αλλά η ακρόαση αυτή είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Εμπορίου, που είναι υπεύθυνη με τον έλεγχο των εξωτερικών, του εξωτερικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται με αυτό το σημαντικό θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Χαίρομαι που οι συνάδελφοι θεώρησαν ότι έπρεπε να γίνει η συζήτηση αυτή στον σωστό και έφθετο χρόνο. Σαν πολιτική οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα θα έλεγα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ομιμότητα των εμπορικών δραστηριοτήτων. Δεν μπορούμε να αγνοούμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τόσα πολλά ζώα και φυτά στον πλανήτη μας. Όχι μόνο έχουμε την υποχρέωση για να διασφαλίσουμε την πολυμορφία αυτή, αλλά έχουμε ευθύνη και στις επόμενες γενιές, γιατί αν δεν πάρουμε δράση, δεν αναλάβουμε συγγνώμη δράση, δεν θα έχουν την ίδια κληρονομιά να φροντίσουν με εμάς. Η κλίμακα εμπορίας ζώων κυρίως από την Άγρια Πανίδα, ειδών από την Άγρια Πανίδα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Όπως βλέπει και η οργάνωση Ελέφαντες Χωρίς Σύνορα in nearly all of uh, sub-Saharan Africa. Τα στοιχεία τα στατιστικά δείχνουν από τη 7 μέχρι 14 ο πληθυσμός των ελεφάντων μειώθηκε κατά 30%, δηλαδή 144.000 ελέφαντες λιγότερο. Ε, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Μοζαμβίκη και η Τανζανία οι εγκληματικές δραστηριότητες έφτασαν σε βιομηχανικό επίπεδο. Στην Τανζανία από 109.000 το 2009 έφτασε στις 43.000 το 2014. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε περίπου για 85.000 νεκρούς ελέφαντες. Στη Μοζαμβίκη 48% αύξηση του αριθμού των νεκρών ελεφάντων πράγματι αυτό είναι χωρίς προηγούμενο. Ένα δεύτερο αρνητικά εντυπωσιακό στοιχείο είναι η αρμόδια υπηρεσία προστασίας της Άγριας Πανίδας των Ηνωμένων Εθνών που ασχολήθηκε με το λαθρεμπόριο των ειδών αυτών, όχι μόνο με τις παράνομες δραστηριότητες, αλλά και με τις δραστηριότητες της εμπορικές που δεν καλύπτονται από τις διεθνείς συμβάσεις. Δυστυχώς ε, η έκθεση αυτή που υπογράφεται από εκπροσώπους 18 χωρών ε, της Αφρικής δείχνουν ότι η εμπορική αυτή δραστηριότητα αντιπροσωπεύει ένα κύκλο εργασιών που φτάνει τα 18 δις σε αιτήσια βάση. Να μην ξεχνάμε λοιπόν ότι η εμπορία των προϊόντων αυτών είναι παράνομη και δυστυχώς μαθαίνουμε πολλά για τα ίδια αυτά, αλλά για τους λάθος λόγους πια, για τη σπανιότητά τους. Και στην Διεθνή Σύμβαση Σάιτες και στο COP17 Έγιναν προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό κατεπηγόντως και θα πρέπει να το διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο προτεραιότητας. Συνεπώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε την πιο πραγματιστική και επίγουσα απάντηση να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των ειδών και να βοηθήσουμε τις επόμενες γενναίες. Θα τελειώσω με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, με μια παρατήρηση θα έλεγα η οποία είναι από τις πιο τραγικές, αν δεν πάρουμε τουλάχιστον μέτρα τώρα. Στις παιδιάδες της κεντρικής Κένια υπάρχει το Old Ketia, ένας χώρος διατήρησης ειδών, και υπάρχουν οι τρεις τελευταίοι βόρειοι λευκοί ρινόκεροι οι οποίοι ζουν από, κάτω από συνεχή φρούρηση ενόπλων. Ε, υποτίθεται ότι κάποιο πρόγραμμα θα μπορούσε χρησιμοποιώντας σαν βάση τα τρία αυτά ζώα να τα αναπτύξει ξανά. Αλλά δυστυχώς οι δύο τελευταίοι ειρηνόκυροι δεν είναι σε θέση να αναπαραχθούν και έτσι λοιπόν αυτά τα τρία περίφημα ζώα θα είναι τα τελευταία του είδους τους μέχρι τη στιγμή τουλάχιστον που αναπόφευκτα θα χαθούν από τον κόσμο αυτό. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν και άλλα ζώα τα οποία θα έχουν την ίδια τύχη. Λοιπόν δεν υπάρχει μια λύση ε, η οποία να είναι μαγική και να βοηθήσει να λυθούν όλα τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να εξετάσουμε την εμπορική μας πολιτική και την τελεμιακή μας πολιτική σαν μια ευκαιρία για την καταπολέμηση των παράνομων εμπορικών δραστηριοτήτων προϊόντων της Άγριας Πανίδας. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλα τα μέσα μας για να θέσουμε ένα τέλος σε αυτό το εμπόριο, το οποίο έχει συνεισφέρει τόσο πολύ στην καταστροφή και χρηματοδοτεί εγκληματικές δραστηριότητες και τρομοκρατία. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω και τις απόψεις των φιλοξενουμένων μας σήμερα Ελπίζουμε να βοηθήσουμε να σταματήσουν αυτές οι πολύ ανησυχητικές εξελίξεις. Thanks Σας ευχαριστώ πολύ που ορίσατε το πλαίσιο της συζήτησής μας. Ξεκινάμε με την πρώτη συνεδρία. Θα ασχοληθούμε με το πλαίσιο πολιτικής, την βιωσιμότητα της Άγριας Πανίδας. Και πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Κούνιο Μικουρίγια, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνίων από το 2009. Και ήδη από το 2014 έχει καλέσει όλες τις ετελωνιακές αρχές να επαγρυπτούν για το πρόβλημα της άγριας πανίδας. Με χαρά θα ακούσουμε τις απόψεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνίων. Κύριε Μικουρίγια, έχετε το λόγο για 8 λεπτά περίπου. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Okay. No, thank you. Technology, it's uh, sometimes... Σας ευχαριστώ. Ε, ξεπεράσαμε τα τεχνολογικά προβλήματα από ό,τι βλέπετε. Ε, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να πάρω το λόγο ενώπιον αρτής της Επιτροπής, γιατί η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας, η εμπορική πολιτική, η σχέση όλων αυτών είναι κάτι που ανησυχεί στη διεθνή κοινότητα. Θέλω να πω δύο λόγια καταρχάς για την Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνίων, η οποία είναι μια διεθνής διακυβερνητική οργάνωση που αποτελείται από τελωνιακέ διοικήσει. Ιδρύθηκε το 1952 στις Βρυξέλλες Και τα πρώτα μέλη της οργάνωσης αυτής ήταν οι τελωνιακές αρχές των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε δηλαδή μία από τις ακρογωνιές λίθους της Ευρωπαϊκής Τελωνιακής Ένωσης. Στη συνέχεια ο φορέας μας έγινε διεθνής και σήμερα έχει 180 μέλη. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των τελωνιακών δραστηριοτήτων και της τελωνιακής διοίκησης, καθορίζοντας πρότυπα και παρέχοντας τεχνική βοήθεια, ε, επίσης ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία. Γνωρίζετε ότι τα τελωνία βρίσκονται πάντοτε στα σύνορα κάθε χώρα σε στρατηγικά σημεία. Ω εκ τούτου, παραδοσιακή λειτουργία των τελωνίων είναι να εισπράττουν εισοδήματα για τα κράτη. Η αποστολή μα όμω έχει εξελιχθεί. Προστατεύουμε την κοινωνία από το λαθρεμπόριο. Καλούμαστε να προωθήσουμε και να διευκολύνουμε το νόμιμο εμπόριο. Επομένως, η εμπορική διευκολύνσεις, η προστασία της κοινωνίας είναι ε, μέρος των καθηκόντων μας. Και για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους αξιοποιούμε τις δυνατότητε τη τεχνολογία για τη διαχείριση κινδύνου στα σύνορα. Σε αυτό το πεδίο της ε, άγριας, πανίδα αυτό που κάνουμε είναι να ε, έχουμε εκστρατείες συνειδητοποίησης. Οι τελωνιακές αρχές ανήκουν στη διοίκηση και πρέπει να θέσουν προτεραιότητες και να ιεραρχήσουν τα περιστατικά. Κάνουμε έρευνα Έχουμε κάνει έρευνα μεταξύ των 180 μελών των 180 τελωνιακών διοικήσεων και πολλές απάντησαν ότι θα ήθελαν να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση του εγκλήματος που συνδέεται με την άγρια πανίδα, αλλά υπάρχει έλλειψη πρώτον νομικού πλαισίου, δεύτερον ανθρώπινων πόρων και τρίτον οικονομικών πόρων. Και αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε. Το 2014 υιοθετήσαμε μία δήλωση μια διακήρυξη για το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας υπογραμμίζοντας ότι η τελωνιακή διοίκηση είναι διαθέσιμη να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί σε αυτό το επίπεδο και η κυβέρνηση, το κράτος, οφείλει να παράσχει περισσότερους πόρους και περισσότερη στήριξη υπό αυτή την έννοια. Επίσης, ζητούμε και τη στήριξη της κοινή γνώμης. Επίσης, γιατί καλούμαστε να λειτουργήσουμε εντός των κοινωνικών πλαισίων και χωρίς τη στήριξη της κοινωνίας είναι δύσκολο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να φέρουμε σε πέρα στα καθήκοντά μας. Με τη... Εάν υπάρχει υποστήριξη από την κοινωνία τότε μπορούμε να έχουμε και πολιτική στήριξη για να φέρουμε σε πέρα στο έργο μας και να μας αυξήσουν τις αρμοδιότητες σε θέματα ερεύνης, ερευνητικά. Διότι πρέπει να μπορούμε να ε, ε, εξετάσουμε και να επιθεωρήσουμε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρέπει να μπορούμε να μεταβούμε εκεί δηλαδή και να έχουμε αυτή την εξουσιοδότηση για να μπορέσουμε να ε, εξουδετερώσουμε αυτά τα δίκτυα τα λαθρεμπορικά. Από εκεί και πέρα, στην υποσαχάρια Αφρική, στις, υποσα... στις χώρες προέλευσης ξεκινήσαμε εν το project Inama. Inama σημαίνει άγρια πανίδα ε, στη γλώσσα της Ζάμπια και με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων χωρών, κυρίως της Σουηδίας, της Γερμανίας, αλλά και χωρών εκτός ΕΕ, όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και με τη στήριξη της γραμματείας του ΣΥΤΕΣ, της Διεθνής Συνθήκης αυτής, εκπαιδεύουμε τους ε, ε, αξιωματούχους για το πώς θα εντοπίζουν καλύτερα τέτοιου είδους φαινόμενα και για το πώς μπορούν να συνεργαστούν με άλλες κρατικές αρχές, με τις αρχές επιβολής του νόμου, για να εξουδετερώσουν τις εγκληματικές αυτές οργανώσεις. Και όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ε, ε, φαίνεται, αυτό από τα ευρήματα της έρευνάς μας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ καλούς πόρους. Άνω του 60% ε, των ευρωπαϊκών τελωνιακών διοικήσεων έχουν διευρεμένη εντολή για τα θέματα αυτά. Όμως οι τελωνιακές αρχές σε πολλές χώρες της Αφρικής δεν έχουν αρμοδιότητα και δεν έχουν και τους σπόρους αλλά δεν έχουν και την κατάρτιση και αυτό προσπαθούμε να το καταπολεμήσουμε. Κάνουμε λοιπόν δράσεις κατάρτισης και μετά την κατάρτιση οργανώνουμε κοινέ δράσεις για να υπάρχει εμπειρία επιτόπου. Πώς μπορεί κανείς να δεσμεύσει αγαθά και πώς να διερευνήσει τέτοιου είδους περιπτώσεις σε συνεργασία με ε, αρχές επιβολής του νόμου αλλά και με ξένες διοκτικές αρχές. Και έρχομαι έτσι ε, σε ένα άλλο πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, το οποίο είναι και η διεθνής εταιρική σχέση. Ε, συνάπτουμε εταιρικές σχέσεις συνεργασίες με άλλους διεθνείς φορείς, θέλουμε να έχουμε συμπράξεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Έχουμε τέτοιου είδου συνεργασίες με το ΣΥΤΕΣ, τη Συνθήκη για την Προστασία της Άγριας Ζωής, με την ε, Europol, με την Interpol, με διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Θα πρέπει τα τελωνία να δουλεύουν χέρι-χέρι με την αστυνομία και τις λοιπές διοκτικές αρχές. Καλλιεργούμε τη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις τις μεταφορικές. Θέλουμε να διευκολύνεται το νόμιμο εμπόριο, να το διευκολύνουμε εμείς και ταυτόχρονα να καταπολεμούμε το λάθρο εμπόριο. Επομένως, η εταιρική σχέση με τους εμπορικούς εταίρους είναι εξαιρετικά σημαντική. Και υπ' αυτή την έννοια έχουμε συστήσει μια task force ενωμένη για την άγρια πανίδα και ε, Φέτος στο Λονδίνο υπεγράφει η δήλωση του Buckingham Palace, όπου ε, όπου δείξαμε στις μεταφορικές ε, εταιρείες ποια ο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να συμμορφούνται όταν ε, να υπάρχει συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις όταν γίνεται νόμιμη μεταφορά άγριας πανίδας και πώ θα καταπολεμούν και θα εντοπίζουν τέτοιου είδου περιστατικά ε, παράνομη μεταφορά άγρια πανίδα. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεργάζονται ε, όλοι όσοι βρίσκονται στα σύνορα, όλο το συνοριακό προσωπικό, όχι μόνο το τελωνιακό. Και έχουμε έτσι υπογράψει μνημόνιο κατανόησης με τους συνεργαζόμενους φορείς, έτσι ώστε να υπάρχει πληροφόρηση, να υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη, να αξιοποιείται όλη αυτή η εμπειρογνωμοσύνη στα σύνορα και να εξουδετερώνεται το λαθρεμπόριο και οι διακινητές. Συμπερασματικά να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερως την διοργάνωση αυτής της ακροάσης γιατί έτσι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη στήριξη και θα διαδώσουμε περισσότερο το μήνυμά μας και έτσι οι εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν αυτό το σκέλος της καταπολέμησης του λαθρομπορίου άγριας πανίδας. Περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στην τελευταία σας ε, πρόταση για τις εμπορικές συμφωνίες που είναι και μια σωστή εισαγωγή για την κυρία Μάντλιν Τουινίγκα που είναι η επικεφαλής της ομάδος της μονάδος D1 εμπόριο και αηφόρος ανάπτυξης της DigiTrade. Ξεκινήσαμε το πρωί με ένα πρόγευμα, με ένα πρωινό για το δίκαιο εμπόριο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γιατί αντιμετωπίσαμε και το θέμα της άγριας πανίδους και σε συνάρτηση με το ελεύθερο εμπόριο, με το δίκαιο εμπόριο μάλλον, και θέλουμε τώρα να δούμε πώς οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να αποτελέσουν και τμήμα του αγώνα κατά του παράνομου εμπορίου. Παρακαλώ. Καλό απόγευμα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτά τα εισαγωγικά σχόλια. Μα μου αρέσει το, το πρωινό με fair trade, αλλά θα προτιμούσα να μην περιέχει το πρωινό μου άγρια πανίδα. Καλύτερα να παραμείνουν ζωντανά αυτά τα άγρια ζώα. Σας ευχαριστώ πάντως για την ευκαιρία να είμαι παρούσα μαζί με τους συναδέλφους μου από την G Περιβάλλοντος. Και αυτό δείχνει τι κοινέ προσπάθειε τη Κομισιόν στον τομέα αυτό. Η Κομισιόν έχει αναγνωρίσει την σοβαρότητα τη τωρινή κατάσταση σε ό,τι αφορά το παράνομο εμπόριο αγρίας πανίδα με το σχέδιο δράση κατά της λαθεμπορίας αγρίων ζώων ξεπερνάει την βασική, το βασικό θεματολόγιο διατήρησης της άγρια ζωή, και περιλαμβάνει πια και τον αγώνα κατά των εγκληματικών οργανώσεων. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ και προσωπικά σε πολλά μέλη του κόσμου και επομένω έχω συνειδητοποιήσει <clears throat> την τροτότητα του οικοσυστήματος από το οποίο κινδυνεύουν να εξαφανιστούν πολλά άγρια ζώα. Η Κομισιόν λοιπόν θέλει να βρει μια σωστή προσέγγιση για να αντιμετωπίσει το λαθρεμπόριο αγρίων ζώων και να προστατεύσει τα ζώα αυτά. Αυτό είναι ένα πολυσχηδές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει αλλαγέ στον έλεγχο των τελωνίων, δημιουργία ικανότητα ε, κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Σάιτος είναι το κύριο εμπόριο με του, του οποίου γίνεται αυτή η ρύθμιση και ο συνάδελφός μου μπορεί να επανέλθει για το θέμα αυτό σε λίγο για το αποτέλεσμα της ε, συνεδρίασης των εμπλεκομένων μερών που περατώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το site του είναι ένα πραγματικό εργαλείο γιατί οι αποφάσεις του επηρεάζουν το εμπόριο άγριας, ε, αγρίων ειδών σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν εμείς ε, διαπραγματευόμαστε για τέτοιες συμφωνίες, η Κομισιόν έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή των πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον, όπως και του άλλου σε τέτοιες συμφωνίες. Θα δείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπόριου για την άγρια ζωή σε διάφορα κεφάλαια των ε, συμφωνιών. Για τις ε, ενεξελίξει ε, διαπραγματεύσεις, αυτό περιλήφθηκε στις διαπραγματεύσεις ticket από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του τους στην Συμφωνία Ελευθερία Εμπορίου με το Βιετνάμ περιλάβαμε και πρόνοιες για μείωση της ε, προσπάθειας για τη μείωση της ζήτησης για προϊόντα άγριας ζωής. Και στον ΠΟΕ η Κομισιόν είναι ενεργό συμμετέχων στην Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος που είναι μια πολύ σημαντική Επιτροπή, κατά την άποψή μα, για να υπάρξουν συνέργειε μεταξύ των δύο αυτών περιοχών. Έχουμε παρουσιάσει μια σειρά από πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί και θα έχουμε σαν στόχο να παρουσιάσουμε στην επόμενη συνεδρίασή τη το σχέδιο για την προστασία τη άγρια ζωή. Πρωτού δώσω το λόγο στον Χαν Στίλστα, τον συναδελφό μου, θέλω να υπογραμμίσω την απόλυτη δέσμευσή μα στο να είμαστε μαζί σα και να... που καταδεικνύεται και από το γεγονό ότι ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε μαζί σα. Ο τρίτος μας ομιλητής λοιπόν θα είναι ο Hans Στίλστα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, είναι επικεφαλής μονάδος για την πολυμερή πολυπεριβαλλοντική συνεργασία. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Και Ευχαριστώ και εγώ από τη δική μου πλευρά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας είναι θετικό το να μπορούμε να ανταλλάσσουμε εμπειρίες από τις προσπάθειές μας. Δύο είναι τα θέματα στα οποία θέλω να σταθώ. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα δράσης. Το ανέφερε ο συνάδελφος. Και δεύτερον είναι οι συμμετέχοντες στη σύμβαση ΣΑΙΤΕΣ, οι ΣΥΤΕΣ σε περιπτώσει. Νομίζουμε ότι η επικοινωνία αυτή είναι κάτι το θετικό για μας. Δυστυχώς δεν έχω πάρα πολλά αντίτυπα για το πρόγραμμα δράσης και δεν θα σας αφήσω το μοναδικό που έχω φέρει άλλωστε. Αλλά έγινε δεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του χρόνου δραστηριοποιούμεθα σε τέτοια θέματα εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι το πρώτο συνολικό πρόγραμμα δράσης το οποίο έχουμε υιοθετήσει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης τον μήνα Ιούνιο και νομίζω ότι και το δικό σας Κοινοβούλιο έχει μπει πλέον στην διαδικασία εξέτασης της πρότασης αυτής, του σχεδίου αυτού, έτσι ώστε να το επικυρώσει με τη δική του σειρά. Υπάρχουν τρεις προτεραιότητες σε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Πρόληψη, πρόληψη των λαθρεμπορικών δραστηριοτήτων. Δεύτερον, δράσεις γύρω από μια πιο αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και σε εθνικό επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο και βοηθώντας τρίτες χώρες να εφαρμόσουν τις νομοθεσίες τις οποίες ήδη έχουν ψηφίσει. Και τέλος, καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων από την Άγρια Πανίδα είναι το πρώτο συνολικό πρόγραμμα δράσης. Εγώ δουλεύω στο τμήμα περιβάλλοντος της Επιτροπής και εμείς ε, έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια αυτή σε συνεργασία και με άλλα τμήματα της Επιτροπής και μετά από διαβουλεύσεις ε, και πέραν του τομέα του περιβάλλοντος, της προστασίας περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε, να φέρουμε σε επαφή όλους τους εμπλεκομένους από τις ΜΚΟ, από τα τελωνία και από άλλους τομείς. Δεν έχω πολλά λεπτά στη διάθεσή μου και γι' αυτό θα σας παρουσιάσω κάποια λίγα στοιχεία από το πρόγραμμα δράσης. Καταρχάς, χρησιμοποιούμε τμήμα της αναπτυξιακής μας συνεργασίας για να υποστηρίξουμε την βελτίωση των δυνατοτήτων που έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να αντιμετωπίσουν τα θέματα της άγριας πανίδας με καλύτερο τρόπο. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα Υπάρχουν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων μία είναι παρούσα εδώ σήμερα και που παρουσιάζουν τις δραστηριότητες τους για την πρόληψη τέτοιων δραστηριοτήτων και τις δυνατότητες που υπάρχουν να αυξηθεί η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να δούμε από κοινού τι μπορούμε να κάνουμε και να υπάρξει καλύτερη νομοθετική ρύθμιση. Υπάρχουν 24 συνολικά δράσεις τις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε, δεν μπορώ να σας τις παρουσιάσω όλες. Ένας άλλος τομέας πάντως έχει σαν στόχο να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την αηφόρο προμήθεια κάποιων υλικών και πρώτων υλών, να υπάρχει σωστή ενημέρωση δηλαδή ότι τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν είναι προϊόντα που προέρχονται από αηφόρες δραστηριότητες. Λοιπόν, αυτά για το πρόγραμμα δράσης. Ένα δεύτερο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω, για μια στιγμή πριν ξεχάσω κιόλας, υπάρχει ένα πενταετές πλαίσιο για το πρόγραμμα δράσης. Ελπίζουμε λοιπόν να το έχουμε πλήρως ε, ολοκληρώσει ε, μέχρι το 2020. Ε, σε αιτήσια βάση θα έχουμε τις λεγόμενες ημέρες της άγριας πανίδας. Και έτσι θα μπορούμε να ελέγχουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος γύρω από τις προτεραιότητες που έχουμε. Τώρα για τη σύμβαση ΣΥΤΕΣ είναι το βασικό διεθνές μέσο για την ρύθμιση του εμπορίου ειδών που βρίσκονται σε κίνδυνο. 183 χώρες συναντώνται κάθε τρία χρόνια και στη συνάντηση την τελευταία που έγινε την προηγούμενες δύο εβδομάδες σημειώθηκε μια μεγάλη προσέλευση ενδιαφερομένων. Η σύμβαση ΣΥΤΕΣ στον τομέα του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερος αποτελεσματική, είναι μία από τις συμβάσεις ιδιαίτερος αποτελεσματικές θα έλεγα. Υπήρξαν 120 πολύ συγκεκριμένες προτάσεις στα πλαίσια της σύμβασης αυτής, η μεγάλη πλειοψηφία έγινε δεκτή αφορά κυρίως μονομενα είδη τα οποία την χάνουν υψηλού ή χαμηλότερου επίπεδου προστασίας. Ταυτόχρονα αφορά και σε κάποιες άλλες προτάσεις έτσι ώστε η διαχείριση της σύμβασης να γίνεται με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Από όλες αυτές τις προτάσεις δεν μπορώ παρά να αναφέρω λίγες Μια πολύ σημαντική πρόταση η οποία έγινε δεκτή και το είχε προτείνει και η Ένωση είναι να υπάρξει μια καταγραφή όλων των ειδών ξύλου ροδόδενδρου. Το rosewood είναι το... η ξυλία από ροδόδενδρο έχει πολύ μεγάλη αξία στην Άπο Ανατολή και λόγω της υψηλής ζήτησης πάρα πολλά είδη ροδόδενδρου ε, βρίσκονται σε κίνδυνο. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να υπάρξει υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ε, μπορεί να γίνουν αντικείμενο εμπορίου ε, μόνο εφόσον έχουν, έχουν υπάρχουν αποδείξεις αν θέλετε ε, για την αηφορία της δραστηριότητας. Τώρα για τον παγκολίνο, ο παγκολίνος είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζώο το οποίο χρησιμοποιείται για παραδοσιακή ιατρική ε, προϊόντα του παγκολίνου βέβαια και λίγες ποσότητες παγκολίνου έχουν ε, φτάσει στην Νοτιοανατολική Ασία τον τελευταίο καιρό και δυστυχώς οι πληθυσμοί παγκολίνου γενικά δεν πάνε καθόλου καλά. Ε, προστατεύεται πλήρως βέβαια το είδος του παγκολίνου, το ίδιο επίσης ε, και τα γκέκο, ηγκουάνα, σάβρες, ε, καρχαρίες, ε, υδράκι του κόμοδου. Γενικά... Thing, because this uh, Νομίζω λοιπόν ότι Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ισχυρό σύστημα το οποίο μπορεί να προστατεύει την άγρια πανίδα και αν κάποιες χώρες δεν εφαρμόζουν σωστά αυτά που προβλέπονται από την σύμβαση υπάρχει επίσης και η δυνατότητα επιβολής πλήρους απαγόρευσης ε, προϊόντων από τα συγκεκριμένα είδη είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέτρο το οποίο θα μπορούσε να ληφθεί και μάλιστα κατά καιρούς λαμβάνεται. Λοιπόν, εδώ θα σταματήσω, Πρόεδρε, γιατί αλλιώς θα ξεπεράσω κατά πολύ το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν το πλαίσιο για την χάραξη πολιτικής Βλέπω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες για να αντιδράσουμε σωστά και να αντιμετωπίσουμε την, σε επίπεδο πλαισίου την λαθρεμπορία. Τώρα, οι συναδελφοί μου έχουν το λόγο για να θέσουν ερωτήματα. Κυρία Φιέλνερ, ένα σύντομα ερώτημα προς την Κομισιόν. Ξέρω ότι η TPP, η Συμφωνία του Ειρηνικού μεταξύ των Πολιτείων και χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας ε, πήρε πολλούς επένους σε σχέση με το κείμενό της για την προστασία το, της άγριας ζωής και για την εφαρμογή των προνοιών του ΣΥΤΕΣ. Και ξέρω επίσης ότι για την πρότασή μας της TTIP έχουμε κάποιες προτάσεις. Ποια είναι η διαφορά μας μεταξύ της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την TTIP σε σχέση με αυτά που συμφωνήθηκαν στην TTP κατά τη συμφωνία του ειρηνικού. Υπάρχουν διαφορές προσέγγισης ή όχι. διαφορέ προσέγγιση Η οχι θα ηταν χρησιμο να ξερουμε ευχαριστω λοιπόν η εμα Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ τους ομιλητές μας. Αν θα μπορούσα να απευθυνθώ στον κύριο Μικουρία για τα τελωνιακά γραφεία. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουν να αντιμετωπίσουν και ποιο ο καλύτερο τρόπο να του βοηθήσουμε. Ποιοι πόροι θα μπορούσαν να του βοηθήσουν να λειτουργήσει καλύτερα η δραστηριότητά του, Και θα μπορούσα να ζητήσω από τους συναδέλφους της DigiTrade αν σε μελλοντικέ συμφωνίες θα περιληφθούν ρήτρε κατά της διαφθοράς και αν θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο. Και αν μπορώ επίσης να ρωτήσω οποιοδήποτε από τους ομιλητές της Κομισιόν για τα αγαθά που είναι σε διέλευση μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή για να ελέγχουμε αυτά τα αγαθά. Και τι είδου πολιτικές υπήρξαν στο παρελθόν μέχρι τώρα αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ντέιβιντ. Καλωσορίζω το γεγονός ότι τον Αύγουστο η Γαλλία απαγόρευσε τελείως το εμπόριο ε, ε, στο κέρας ελέφαντα και ρινόκερου. Αυτό όμως συνάδει με την ενιαία αγορά. Είναι ασυνήθιστο να υιοθετεί μονομερή δράση μια χώρα. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο ευρωπαϊκής απαγόρευσης σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια για να συμπληρώσουμε αυτή τη δράση. Και η Επιτροπή μας ζήτησε να υπάρχει στήριξη για τη συμπερίληψη των Αφρικανικών ελεφάντων στο πρώτο παράρτημα της σύμβασης ΣΥΤΕΣ, της ΆΙΤΕΣ. Τελικά δεν έγινε αυτό. Γιατί όμως. Ο Πρόεδρος και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για τους πόρους των τελωνιακών διοικήσεων. Χθες Κάναμε μία επίσκεψη και συζητήσαμε και με τελωνιακούς για το τελωνιακό κώδικα, για την Αγρία Πανίδα, για την τήρηση του IPR. Πάρα πολλά τα καθήκοντα για την τελωνιακή μονάδα που ασχολείται με τους δασμούς. Ποια είναι η άποψή σας για τους πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε ότι σε ορισμένα μέρη ένα τελωνιακό, για παράδειγμα, είναι υπεύθυνο για 12.000 παιχνίδια που εισάγονται και σε άλλο λιμάνι ένα τελωνιακό είναι υπεύθυνο για 36.000 παιχνίδια. Όταν έχουμε τόσα πολλά κοντέινερ που έρχονται στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Είναι πραγματικά δυνατό να εντοπίσει κανείς και να καταπολεμήσει το λαθρομπόριο άγριας πανίδας. Ίσως να ξεκινήσουμε με εσάς κύριε Μικουρίγια. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τις ερωτήσεις σας. Να σας πω το εξής κύριε Πρόεδρε, η τελωνιακή μεθοδολογία είναι η εξής. Υπάρχουν χιλιάδες ε, ε, κοντέινερ και δεν υπάρχουν πόροι να τα ανοίξουμε ένα προς ένα και να δούμε τι έχει το καθένα μέσα. Το σημαντικό είναι η μέθοδος διαχείρισης κινδύνου. Κάθε φορτίο συνοδεύεται από εμπορικά δεδομένα και τα τελωνία λαμβάνουν τα εμπορικά δεδομένα από πριν, ιδανικά από πριν, και εάν τα έχουν λάβει από πριν, τότε μπορούν να τα αναλύσουν Αναλόγως με την προέλευση του φορτίου, ποιος το υπογράφει, ποιος το στέλνει, ποια διασάφηση γίνεται. Έτσι μπορεί να εντοπίσουμε τα ύποπτα κοντέινερ, τα ύποπτα εμπορευματοκιβώτια και μετά έχουμε σκάνερ, έχουμε διάφορα τεχνολογικά μέσα που μας βοηθούν να εντοπίσουμε πραγματικές απειλές. Και όταν όλα αυτά φέρουν ένα αποτέλεσμα, τότε λέμε ότι αυτό το κοντέινερ θα το ανοίξουμε και θα το επιθεωρήσουμε να δούμε τι έχει μέση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν μας βοηθάει, γιατί όλο και πιο μικρά πακέτα φτάνουν στα σύνορα. Και γι' αυτό θέλουμε η βιομηχανία και τα, ε, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να μας στέλνουν περισσότερες πληροφορίες εκ των προτέρων. Αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον. Και ως προς τις προκλήσεις, να σας πω το εξής. Θα πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει το νομικό, με το νομικό πλαίσιο και τους πόρους. Δηλαδή να αλλάξει το νομικό πλαίσιο, να αυξηθούν οι πόροι για να δείξουν οι κυβερνήσεις ότι το θέμα το ιεραρχούν αρκετά ψηλά στην ημερησία τους διάταξη. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεργαστούν οι διοικήσεις μεταξύ χωρών προέλευσης και χωρών ε, παραλαβής ε, σε αυτό το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας για την καλύτερη καταπολέμησή του. Σίγουρα εκεί που ξεκινάει αυτή η αλυσίδα πρέπει να δράσουμε γιατί τα τελωνία αυτή τη στιγμή χάνουν εισοδήματα. Εξετάζουν όμως και τώρα και τις εξαγωγές γιατί συνειδητοποιούν ότι ε, ε, είναι επιβλαβές το λαθρεμπόριο όχι μόνο από την οικονομική σκοπιά αλλά και από την κοινωνική σκοπιά. Έχουμε μια κάποια χρηματοδότηση, ειδικότερα από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένε Πολιτείε και ε, τη διεθνή κοινωνία των μελών μας. Ωστόσο, δίνουμε πόρους για τους τελωνιακούς υπαλλήλους επιτόπου και χρειάζεται εκεί στήριξη έτσι ώστε να συνεργαστούν με τις αστυνομικές, με τις διοκτικές αρχές για να υπάρχει ένα δίκτυο ε, επιβολής του νόμου. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εάν υπάρξουν πόροι από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και από δωρητές στις τελωνιακές αρχές, αυτά θα βοηθήσουν πολύ την καταπολέμηση του ελευθερμπορίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, η Μάτλιν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω απατώντας το πρώτο ερώτημα για την TTIP και την Συμφωνία του Ειρηνικού, TTP. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια πολύπλευρη, αν θέλετε, αντιμετώπιση ενώ άλλες χώρες όπως το Ηνωμένε Πολιτείε απλά εφαρμόζουν την εσωτερική τους νομοθεσία. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να κάνουμε στα πλαίσια και του TTIP βασίζεται στους ΣΥΤΕΣ. στην ουσία υπάρχει μια αμοιβεοποίηση, αν θέλετε, των διαφορετικών νομικών πλαισίων. Αυτό είναι ένα κομμάτι των συζητήσεων που έχουμε γύρω από το TTIP. για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν ασχολούμαι εγώ ίδια άμεσα με τα θέματα αυτά, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν είναι μυστικό ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί ευαισθησία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξετάζεται το θέμα αυτό σε εσωτερικό επίπεδο. Θα συνεχίσω με κάποιες από τις άλλες ερωτήσεις. Κάποιος από σας αναφέρθηκε στην γαλλική απόφαση να σταματήσει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξαγωγή ελεφαντόδοντος. Και η Ολλανδία έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει το ίδιο πράγμα. Και στις δύο περιπτώσεις ενημερώσαμε τις συγκεκριμένες χώρες ότι μπορούν να το κάνουν στα πλαίσια των κοινοτικών νομικών ρυθμίσεων. Θα δούμε πώς θα τεκμηριώσουμε την απάντησή μας προς τις χώρες αυτές βασική μας αντίδραση στην αρχή ήταν να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται βέβαια στην εσωτερική αγορά. Αλλά παρόλα αυτά στα πλαίσια του προγράμματος δράσης μέχρι το τέλος του χρόνου θα προχωρήσουμε στην απαγόρευση εξαγωγών ελεφαντόδοντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς άλλες χώρες, κυρίως την Κίνα. Αλλά αυτό θα ισχύσει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ε, μια ειδική δυνατότητα που μας παρέχει η νομοθεσία για την Άγρια Πανίδα. Είχαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις να αντιμετωπίσουμε όπως το κέρας των ρινοκέρων. Ε, αυτά για τις συζητήσεις με την Γαλλία και την Ολλανδία. Για τις Αφρικανούς ελέφαντες. Έγινε μια τεράστια συζήτηση στο Τζοχάνεσμπεργκ, στην COP17. Η βασική ιδέα η οποία είχε τεθεί ήταν ότι 28 αφρικανικές χώρες που είχαν αφρικανικούς ελέφαντες, που ήθελαν όλους τους ελέφαντες να εντάσσονται στο υψηλότατο επίπεδο προστασίας, το επίπεδο 1 του ΣΥΤΕΣ. Υπήρξαν και κάποιες άλλες χώρες οι οποίες διαφωνούσαν, μια μικρότερη ομάδα χωρών, η οποία όμως ε, μικρότερη ομάδα χωρών έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό ελεφάντων. Αυτή είναι μια παραδική συζήτηση στο ΣΥΤΕΣ και επαναλήφθηκε με πολλές ε, μικιό να υποστηρίζουν τις πολλές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστήριξε την πρόταση αυτή. 71 χώρες στο τέλος καταψήφισαν την πρόταση για την αναβάθμιση των περιορισμών στην εμπορία. Για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι γιατί θεωρήσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα βοηθούσε τους ελέφαντες, δεν θα συνιστούσε έναν αποτελεσματικότερο τρόπο ε, προστασίας από τους λαθροκυνηγούς και θα ήταν και αντιπαραγωγικό διότι αυτή τη στιγμή αποφασίσεις να αλλάξει την ταξινόμηση στα πλαίσια του ΣΥΤΕΣ από το παράρτημα 1 στο 2 αυτό σημαίνει ότι οι χώρες της, του παραρτήματος 2 μπορούν να υπογράψουν μια επιφύλαξη και για να το πω κάπως ε, απλά θα καθιστούσαν ε, άκυρη την αναβάθμιση και θα μπορούσαν να νομιμοποιήσουν έτσι παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε έτσι ώστε να υπερασπιστούμε την πρόταση αυτή για την μη στήριξη της πρότασης από πλευράς των Αφρικανικών χωρών και στο τέλος η πλειοψηφία στα ΣΥΤΕΣ απέρριψε την πρόταση αυτή των 28 Αφρικανικών χωρών. Τέλος, για τα διαμετακομιζόμενα προϊόντα ε, και για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν σημείο διαμετακόμισης ε, προϊόντων λαθρεμπορίου από άγρια ζώα. Η συζήτηση εδώ είναι αρκετά περίπλοκη. Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, αυτό που πρέπει να πω ότι ένας από τους λόγους ε, που ακολουθήσαμε, την στάση που ακολουθήσαμε, είναι γιατί είμαστε σημείο διαμετακόμισης. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η τύχη των Βιετναμέζων κυνηγών που έχουν ε, τσεχική υπηκότητα, που πηγαίνουν στην Νότια Αφρική, κυνηγούν ρινοκαίους, τους φέρνουν στην Τσεχία σαν σαν ε, είναι πανάκριβη η τιμή ε, των αγαθών αυτών, έχει αντίστοιχο κόστος με το χρυσό ή με την κοκαΐνη και μετά τα επανεξάγουν από την Τσεχία στο Βιετνάμ και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πρακτικών που δεν θέλουμε να επαναληφθούν. Και θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την δραστηριότητα. Ένα άλλο θέμα, μια άλλη περίπτωση, είναι ότι όταν ορισμένα αγαθά ε, φτάνουν στους ευρωπαϊκούς λιμένες, οι λιμενικές αρχές ε, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να σταματούν αυτού του είδους τα προϊόντα. Κάποιοι λιμένες στη Βόρεια Ευρώπη ήθελαν να σταματήσει, σαν παράδειγμα, με δική τους πρωτοβουλία η εμπορία κρέατος φάλαινας. Και τελικά είχαμε αποφασίσει ότι οι λιμενικές αυτές αρχές θα πρέπει να είχαν την δυνατότητα να το κάνουν. Και ότι δεν υπήρχε κάτι το παράνομο εκεί σε επίπεδο κοινοτικό. Δεν έχουν κλείσει όμως οι υποθέσεις αυτές. Άλλο παράδειγμα, το οποίο αν ενθυμούμε καλά, χθες το διάβασα, το κοίταξα, ένα πλοίο με σημαία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέφερε από την Ισλανδία στην Ιαπωνία κρέας φάλαινας. Αν περνούσε από τα κοινοτικά ύδατα αυτό θα ήταν παραβίαση της οδηγίας Habitats. Αλλά μετέφερε το κρέας αυτό από το Reykjavik στην Ιαπωνία κάπου και δυστυχώς η υπόθεση αυτή είναι πολύ περίπλοκη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια κάποια δόση ευθύνη εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως και να έχει κάποια μέσα να σταματήσουν οι εμπορικές αυτές δραστηριότητες, αλλά όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση. Yes, uh, thanks a lot. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο ε, πάνελ για την εφαρμογή των μέτρων και εδώ έχω τέσσερις ε, διακεκριμένους ομιλητές. Ο κυρία Γουέν Φόγκ Ντούγκ από το Βιετνάμ, η αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλον, και του Φορέα Προστασίας της Άγριας Ζωής και έρχεται πράγματι από το Βιετνάμ σε αυτή την συνεδρίαση και θα σας δώσω μέσα στο λόγο. Καλημέρα σε όλους. Με ακούτε? Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία να έρθω ενώπιόν σας και να σας εξηγήσω το έργο μας στο Βιετνάμ. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το λαθρεμπόριο αγρίας πανίδος στο Βιετνάμ. Έχω έρθει από πολύ μακριά, από το Χανόι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μάτιο αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα κατά των αγρίων ειδών. Να σας παρουσιάσω το φορέα μας. Εργάζομαι για μια τοπική ΜΚΟ που λέγεται Παιδεία για τους πολίτες του Βιετνάμ. Και είμαστε η πρώτη τέτοια οργάνωση στο Βιετνάμ σήμερα. Όπως ξέρετε το Βιετνάμ έχει υπογράψει πολλές συμβάσεις σε σχέση με τα θέματα των γυναικών και υπάρχει και μια συμφωνία με την ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να εφαρμόσουμε την Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με τις ΗΠΑ, αλλά εμεί ω φορείς διατήρησης των φυσικών πόρων βλέπουμε εδώ και ένα αποτελεσματικό εργαλείο για να προωθήσουμε το θεματολόγιο προστασίας των αγρίων ειδών στο Βιετνάμ και να αντιμετωπίσουμε την παράνομη λαθεμπορία αγρίων ειδών. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα προέρχονται πολλές αλλαγές στο Βιετνάμ για τα θέματα προστασίας. Από ό,τι βλέπετε από τη διαφάνεια υπάρχει και η θέληση των καταναλωτών να ενισχυθεί αυτό το πλαίσιο. Σας δίνω λοιπόν μια επισκόπηση για τα θέματα αυτά. τη δράση μας στο Βιετνάμ. Βλέπετε από αυτή τη διαφάνεια έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για να εργαστούμε και μας έχει βοηθήσει και το Ταμείο Άγριας Πανίδας του ΟΗΕ. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από ενέργειες για να αντιμετωπίσουμε τι ανάγκε των αγρίων ειδών που βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο. Δεν θα πω σε λεπτομέρειε για το πώ το Βιετνάμ έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει το παράνομο λαθρεμπόριο για, τις, ε, για τα άγρια είδη. Κάποιοι από εσά ξέρετε ότι κάποιε από τι πιο μεγάλε υποθέσει για τα θέματα αυτά έγιναν <coughs> στα ε, στο Χανόι και στην πόλη του Χοτσιμίνγκ, όπου υπήρξε κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων αγρίων ειδών. Είναι λοιπόν ένα σημαντικός όγκος ελεφαντόδων του, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτό το λαθρεμπόριο. Είναι η ίδια κατάσταση με τον Παγκολίνο. Το Βιετνάμ δεν είναι μονάχα ένα, μια χώρα τελικού, τελικής κατανάλωσης και μια χώρα διέλευσης έρχονται από διάφορες ε, γειτονικέ χώρες παγκολίνο και το ίδιο συμβαίνει και με τίγρης. Δεν ξέρω αν βλέπετε εδώ πέρα στη διαφάνεια. Έρχονται διάφορα είδη Και πολλές φορές αυτά τα άγρια είδη καταλήγουν στην κατσαρόλα στο Βιετνάμ. Ε, το κρέας από αυτά τα άγρια ζώα είναι πολλά πράγματα λοιπόν πρέπει να κάνουμε στο Βιετνάμ. Είμαστε καταναλωτές αυτών των προϊόντων, είμαστε σημαντική χώρα διέλευσης. Και πρέπει να πω ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, είναι πολλά άτομα τα οποία εμπλέκονται στο εμπόριο αυτό. Η κυβέρνηση του Βιετνάμ δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό για να εξαλείψει αυτό το πρόβλημα. Οι γνώσεις μας από το θέμα αυτό, γιατί εργαζόμαστε εδώ και 10 χρόνια για το θέμα αυτό, <clears throat> αναγνωρίζουμε ότι το Βιετνάμ έχει κάνει σημαντική βελτίωση στα θέματα εφαρμογής Αλλά αυτό το οποίο γίνεται είναι σε νομοθετικό επίπεδο υπάρχουν ε, νέες εγκύκλοι και οδηγίες και έχουμε ένα νέο ποινικό δικαστήριο για τα θέματα αυτά το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί εφέτος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν λάβει χώρα στο Βιετνάμ. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η προσαρμογή της νομοθεσίας στα θέματα αυτά. Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι ιδιοκτικοί φορείς στο θέμα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν οι ανάγκες εφαρμογής του νόμου που δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι οι διαδικασίες δίωξης οι αρχές οι ιδιοκτικές όταν συλλαμβάνουν κάποιο επαυτοφόρο έχουν πολλές δυσκολίες να φέρουν σε πέρας όλη αυτή τη διαδικασία γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν εγκληματικά δίκτυα τα οποία κρύπτονται πίσω από μια τέτοια πράξη και δεν είναι πάντα εύκολο να βρουν αυτούς οι οποίοι έχουν ξεκινήσει αυτές τις διαδικασίες. Είναι λοιπόν μεγάλη δυσκολία για μας η εφαρμογή του νόμου. Βλέπετε εδώ την εμπορία θαλασσινών χελωνών στις, ε, στο Βιετνάμ. Έχουμε πολλές φορές όμως τις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες απειλούν τους μάρτυρες και κανείς δεν θέλει να δώσει πληροφορίες για το θέμα αυτό. είναι ένα μεγάλο μέρος του λαθρεμπορίου, το λαθρεμπόριο στις ε, θαλάσσιες χελώνες. Υπάρχει ένας μεγάλος εγκληματίας επικεφαλής ενός δικτύου, ο οποίος είναι υπό ανάκριση, αλλά δεν έχει ακόμα ε, μπει στην φυλακή και είναι μια ουσιαστική, μια ουσιαστική περίπτωση αυτή για να αποδείξει και η κυβέρνηση του Βιετνάμ ότι μπορεί πράγματι να αντιμετωπίσει αυτό το έγκλημα και τους οργανωτές αυτού του εγκλήματος. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί στο Βιετνάμ είναι να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε την παράνομη εκτροφή ειδών που είναι σε κίνδυνο. Βλέπετε εδώ πέρα τους κροκόδιλους. Πολλοί πιστεύουν ότι μπορεί η εκτροφή κροκοδίλων να είναι μια σημαντική ε, πηγή διατήρησης αυτών των ειδών. Και αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πολλές φορές δεν συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η περίπτωση των ε, τίγρεων. ο κύριος Τουάν έχει ένα αγρόκτημα όπου έχει το δικαίωμα να κρατάει τίγρης για σκοπούς προστασίας των αγρίων ειδών. Αλλά αν δώσετε αυτή την ευκαιρία μπορεί να υπάρξει εμπόριο τίγρεων. Έτσι έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν ζωντανές τίγρης στα αγροκτήματά του. Αυτό είναι ένα θέμα που κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να μην ξέρουν για ποιο λόγο πηγαίνουν οι τίγρες εκεί πέρα και στέλνουν τις τίγρες στο Βιετνάμ που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το εμπόριο. Έχουμε το θέμα της, εμπο... της ε, ε, εταιρικής κοινωνικής ασφάλειας, συγγνώμη, ευθύνης, δεν αναφέρεται τίποτα στην ε, ε, συζήτηση για τα θέματα αυτά στο Βιετνάμ είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν, να εμπλέξουν αυτήν την ε, ευθύνη των επιχειρήσεων για την προστασία της άγριας ζωής. Έχουμε λοιπόν πολλά τέτοια είδη. Υπάρχουν πολλές δυτικές εταιρείες και μεγάλες εταιρείες οι οποίες είναι πάντα έτοιμες να εκμεταλλευτούν τα ίδια αυτά στην παραγωγή των ε, ειδών τα οποία θέλουν στην αγορά. Χρησιμοποιούν ενδιάμεσες εταιρείες στο Βιετνάμ και δεν υπάρχει η ικανότητα να παρακολουθηθεί όλος αυτός ο κύκλος. και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παρανόμων ειδών. Έχουμε λοιπόν <clears throat> πάρα πολλά εμπόδια, αλλά συγχρόνως υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες σήμερα στο Βιετνάμ να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να έχουμε καλύτερη προστασία των αγριών ειδών. Έχουμε ένα νέο νόμο ένα νόμο περί ιδιοκτησίας, ο οποίος αφορά και την ανάγκη να υπάρχουν επίσημοι τίτλοι για την ε, ιδιοκτησία γης. Αυτό θα βοηθήσει την προστασία της άγριας ζωής. Έχουμε επίσης, όπως το είπα προηγουμένως, και ένα νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή εφέτος, δηλαδή το 2017. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει καλύτερος κολλασμός των παραβατών. και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες επίσης και με το EVFTA. Γιατί εκεί υπάρχει έμφαση στην ε, εφαρμογή της νομοθεσίας για, τις, ε, για την άγρια πανίδα και επίσης οι πολυμερείς συμφωνίες, παραγωγός χάρη εκτροφή τίγρεων. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πλαίσιο ρύθμισης το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει. Ένα άλλο σύντημα το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η πρόθεση της εταιρική ευθύνης στο Βιετνάμ και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, τοπικών NGOs, των τοπικών μη κυβερνητικών οργανώσεων, ώστε να συνεχιστεί η παρακολούθηση της δυνατής ε, παραβίασης της νομοθεσίας για την Αγρία Πανίδα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Overview about the situation in Vietnam. Our next speaker is... Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κάουτσμαν της DHL. Signed the United for Wildlife Transport Task Force η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και θα μας πει πώς βοηθά την καταπολέμηση της δραστηριότητας αυτή. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, λέει ο κ. Κάουτσμεν. Το πρόβλημα έχει παρουσιαστεί με σωστό τρόπο από τους προηγούμενους ομιλητές. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση, πολύ κρίσιμη αυτή που έχει δημιουργηθεί. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις εμπειρίες τις οποίες είχα εγώ συνεργαζόμενος με κάποιες από τις ε, πρωτοβουλίες και τις ομάδες τις οποίες αναφερθήκατε ήδη και οι οποίες νομίζω ότι βοήθησαν τα πράγματα να βελτιωθούν κάπως. Καταρχάς θεωρώ ότι η πρόθεση, η επιθυμία να βοηθήσει κανείς προς την κατεύθυνση αυτή και το πάθος είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τη δράση μας και το λέω αυτό παντού και το βλέπω παντού. Είναι μακρύς ο δρόμος βέβαια τον οποίο θα πρέπει να διανύσουμε και θα φανεί αν πράγματι μπορούμε να επηρεάσουμε τα πράγματα. Πολλοί εμπειρογνώμονες είναι απεσιόδοξοι, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην συνεχίσουμε την προσπάθεια. Υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές πρωτοβουλίες και κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις εγώ ασχολήθηκα με το Ίδρυμα Τάσκ στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως επίσης και με το Ίδρυμα George Άνταμ στην Τανζανία, που προσπαθεί να ξαναφτιάξει ένα μεγάλο πάρκο προστασίας, όπως επίσης και το πάρκο Μποκανάζη στη Βόρεια ε, Τανζανία. Οι άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες έχω εμπλακεί προσωπικά είναι το United for Wildlife από το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 1,5 χρόνο. Το United for Wildlife είναι θα έλεγα σαν μια οργάνωση υποδειγματική γιατί ξεκίνησε από μια συγκεκριμένη προσπάθεια έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στον τομέα των μεταφορών των ειδών αυτών. Είχαμε λοιπόν μια συγκεκριμένη εντολή αν θέλετε, ε, κράτησε κάτι παραπάνω από το χρόνο που είχαμε προβλέψει, αλλά κατάφερε να συνδυάσει ισχυρούς παίκτες της βιομηχανίας και τον πρόεδρο της ΙΑΤΑ, επίσης τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ματζέλαν, εγώ που εκπροσωπώ το ε, το DHL, την Maersk ε, και γενικά και άλλες επιχειρήσεις και ΜΚΟ. Και νομίζω ότι ε, είχαμε πολλά να κερδίσουμε από την παρουσία επίσης εμπειρογνωμόνων και από τα Τελωνία, την Μέση Ανατολή και την Ιαπωνία. Νομίζω λοιπόν ότι υπογράψαμε όλοι μια πολιτική που θα χαρακτήριζα μηδενικής ανοχής για τη μεταφορά των ζώων αυτών, κάτι το οποίο ήταν έτσι και αλλιώ μια θα έλεγα ένα βασικό επίτευγμα. Ένα άλλο επίτευγμα σημαντικό είναι το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο ε, θα έλεγα χρησιμοποιείται για την ε, κυκλοφορία των πληροφοριών αυτών, κάτι το οποίο δεν γίνεται με διαφορετικό τρόπο, ε, ούτε καν σε επίπεδο τελωνιακών αρχών. Η δική μου εταιρεία έχει βοηθήσει στην προσπάθεια αυτή και νομίζω ότι κάναμε κάτι το οποίο ε, μπορεί να εντοπιστεί με συγκεκριμένο τρόπο Εμείς στην ουσία καταγράψαμε αν θέλετε όλες τις ε, προσπάθειες που κάνει το United for Wildlife σε όλους τους εργαζομένους μας στον κόσμο, 700.000 περίπου. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν ε, τις προσπάθειες αυτές και με τα εσωτερικά μέσα ενημέρωσης και με τη σωστή κατάρτιση και ε, στην ουσία ενσωματώσαμε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στοιχεία από το θέμα αυτό. Είναι κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν είχε απασχολήσει πολύ και υποθέτω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντικατοπτριστεί σύντομα και σε άλλες δραστηριότητες των τομέα των μεταφορών και του ελέγχου. Ο έλεγχος στην δική μας περίπτωση, όπως είπε και η προηγούμενη συνάδελφος, είπε το, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς ε, κάθε ε, εμπορευματοκιβώτιο. Υπάρχουν όμως κάποιοι τρόποι, υπάρχουν κάποιες μέθοδοι και εταιρείε, υπάρχουν ε, επίσης και έλεγχοι τυχαίοι θα έλεγα, αλλά τακτικοί των εμπορευματοκιβωτίων σε διαμετακόμιση αλλά ιδιαίτερα στις αερομεταφορές μπορεί να γίνουν περισσότερα και σε ακτίνες ε, χ, ε, αυτές που χρησιμοποιούνται για να ελέγχονται ε, τα, οι τσάντες και των επιβατών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει και η δική μας πλευρά να επενδύσει περισσότερο εδώ και αυτό θα είναι αποτελεσματικό μακροπρόθεσμα. Η τρίτη δράση την οποία έχουμε αναλάβει είναι να προσπαθήσουμε να μετακινούνται κάποια ζώα και γι' αυτό δωρήσαμε τη χρήση ενός αεροσκάφους, μεταφέραμε από το Κέντ τρεις ρινόκερους ε, στο καταφύγιο Μοκαμάζη της Βόρειας Τανζανίας Ε, δύο από αυτούς γέννησαν ε, νέα ζώα ε, μετά από δύο χρόνια και το πρόγραμμα λοιπόν αναπαραγωγής δούλεψε ενώ στο παρελθόν ήταν η κατάσταση απελπιστική. Μεταφέραμε επίσης και μια μεγάλη οικογένεια από γορίλες στο Κονγκό, στο σπίτι τους. Και αυτό το κάναμε σε ένα περιβάλλον πιο ανοιχτό βέβαια μεταφέραμε τίγρης ε, από την Αυστραλία, μια τίγρη από το Οχάιο και τους βάλαμε σε καλύτερο περιβάλλον στο Λονδίνο. Εγώ δεν ζητάω να μου πείτε τι καλά που τα κάνατε, αλλά να σας δείξω ότι μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα από την εταιρεία μεταφορών εάν υπάρχει πάθος. Λόγω ακριβώς αυτής της συνειδητοποίησης ε, του προβλήματος βρίσκουμε περισσότερα παράνομα ε, είδη, ερπετά, πουλιά και σε, μικρά, σε μικρές βαλίτσες και αποσκευές ακόμα. Λοιπόν, είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα εδώ να πω είναι ότι συντονίζοντας την δράση μας με όλους τους εμπλεκόμενους και που ενδιαφέρονται για αυτά, όπως το United for Wildlife, αν μπορέσουμε λοιπόν να συνδυάσουμε τις προσπάθειες και αν μπορέσουμε να συνδυάσουμε την εμπειρογνωμοσύνη όλων, τότε μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά τα πράγματα. Και πράγματι αυτό νομίζω είναι το βασικό σημείο, η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανταλλαγή γνώσης. Γιατί αν δεν υπάρξει συνέχιση της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει, τότε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικά διάστημα δεν θα γίνεται τίποτα και συγχαίρω τους προηγούμενους ομιλητές για την αποφασιστικότητα και το πάθος το οποίο επέδειξαν. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι η Μισελ Όουεν. που θα αποεπροσωπεί ένα διεθνές δίκτυο παρακολούθησης της Άγριας Πανίδας, μία από τις πιο σημαντικές ΜΚΟ σε αυτό το τομέα. Έχετε το λόγο κυρία Όουεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις ε, για το τράφικ. Έτσι γλιτώνω χρόνο. Είμαστε μία μήκη που εξετάζει το εμπόριο και το νόμιμο εμπόριο και το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας. Εδώ είναι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και γι' αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το εμπόριο άγριας πανίδας μπορεί να είναι νόμιμο Όλοι εποφελούμαστε από αυτό γιατί από αυτό προκύπτουν έπιπλα ρούχα τρόφιμα και αποτελεί και πηγή πλούτου εισοδήματος για πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Αυτό αναφέρεται και στη σύμβαση ΣΥΤΕΣ, ε, τη σύμβαση που ελέγχει το νόμιμο εμπόριο άγριας χλωρίδας και πανίδας. Υπάρχουν προαπαιτούμενα σε αυτή τη σύνδεση που, σύμβαση που ελέγχουν το νόμιμο εμπόριο πάνω από 35.000 ήδη απαριθμούνται και υπάρχει προαπαιτούμενο να υπάρχει άδεια για εισαγωγή, εξαγωγή και επανεξαγωγή τέτοιου είδους, ε, για τέτοια είδη. Οι άδειε αυτές πολύ συχνά αναπαράγονται ή πλαστογραφούνται, παραποιούνται, ε, το υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης είναι το εσφαλμένο και αυτά είναι τα προβλήματα όταν προσπαθεί κάποιος να προλάβει έτσι ώστε το νόμιμο εμπορικό σύστημα να μην το αξιοποιούν τα παράνομα κυκλώματα. Τώρα το λάθρεμπόριο είναι μία από τις πιο μεγάλες εγκληματικές αγορές στο κόσμο. Οι αξίες ποικίλουν, αλλά γενικά η αξία αυτής της αγοράς είναι άνω των 20 δις δολαρίων ετησίως. Και την αγορά αυτή νέμονται οργανωμένα ε, εγκληματικά δίκτυα και έχουμε εμβληματικά ήδη έχουμε κυρίως το ελεφαντόδοντο, το ελεφαντοστούν και το καθεξής, αλλά έχουμε και ε, λαθρεμπόριο μεταξύ Αφρικής Ασίας, μεταξύ εντός της ίδιας Ασίας, αλλά έχουμε και λαθρεμπόριο με είδη που έρχονται από την Νότια Αμερική. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το μέγεθος του προβλήματος και το ότι συνδέεται αυτό το λαθρομπόριο με τις εγκληματικές οργανώσεις. Αυτό το έχουν παράξει πολλές κυβερνήσεις και γι' αυτό έχουν αναλάβει δεσμεύσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια οι ΙΠΑ έχουν εθνική στρατηγική με τοπικά και διεθνή χαρακτηριστικά. Οι 41 χώρες που έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν την, το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας το έχουν κάνει με τη δήλωση του Καζάνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέδιο δράση σχετικό. Αναφέρθηκε και η δήλωση του Μπάκιν Χαμπάλας, ενωμένη για την άγρια ε, πανίδα. Ε, φαίνεται δηλαδή ότι όλο και περισσότερο εμπλεκόμενοι φορείς θέλουν να αναλάβουν και αναλαμβάνουν δράση. Τον Απρίλιο αυτής της χρονιάς η ΑΙΑΤΑ ενέκρινε ομόφωνα ένα ψήφισμα ε, που έχει μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου κατά την αεροπορική μεταφορά στο τράφικ σε αυτό το δίκτυο. Εγώ είμαι επικεφαλής ε, μιας εταιρική σχέσης που αποτελείται από διοικητικούς, δημόσιους και ιδιωτικού φορείς έτσι ώστε να μειωθούν οι δυνατότητες που έχουν οι λαθρέμποροι διακινητές να αξιοποιήσουν τις νόμιμες οδούς του εμπορίου. Στηρίζουμε τον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση των συστημάτων τους. Εξετάζουμε πώς μπορούμε να του δώσουμε στοιχεία, πληροφορίες στον ιδιωτικό τομέα για να βελτιώσει τα συστήματά του. Ε, συνεργαζόμαστε με τους επικεφαλείς των εταιριών έτσι ώστε να υπάρχει εμπιστασύνη και αλληλοϊποστήριξη. Δίνουμε εκπαίδευση, κατάρτιση έτσι ώστε να έχουν τις δυνατότητες οι εταιρείες να εντοπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα εξετάζουμε από κοινού με τις εταιρείες την πολιτική τους, πώς μπορούν να την αναθεωρήσουν και προσπαθούμε να ε, αυξήσουμε τις γνώσεις και τη συνειδητοποίηση αυτού του προβλήματος. Δεν ε, ασχολούμαστε με τις διοκτικές αρχές. Ε, βοηθούμε τις ιδιωτικές εταιρείες που δεν έχουν αρμοδιότητα στην επιβολή του νόμου. Εάν δείτε την αλυσίδα εφοδιασμού και μεταφοράς, καταλαβαίνετε ότι η εφαρμογή όλων αυτών είναι τεράστια πρόκληση. Είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα, πάρα πολλέ οι χώρε από τι οποίε διέρχεται η μεταφορά, Εμπλέκεται η αστυνομία, η τελωνιακή διοίκηση, οι μεταφορεί, οι ιδιωτικέ εταιρείε, πάρα πολλοί φορεί που δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολή του νόμου. Α πάρουμε ένα παράδειγμα αεροπορική μεταφορά. λαθρεμπόριο, δηλαδή άγρια σπανία μέσω αυτού του συστήματο. Ένα επιβάτης μπορεί να το κάνει με πολλού διαφορετικού τρόπου. Μπορεί να το βάλει σε αποσκευέ του, να το μεταφέρει πάνω του, να το στείλει όσο φορτίο για να αποφύγει την ανείχνευση, τον εντοπισμό. Αυτή η κυρία προσπαθούσε να φέρει αυγά και προσπαθούσε να αποφύγει την ανείχνευση από τα σκάνερ. Βλέπετε πόσο φυσιολογικά φαίνονται όλα στη φωτογραφία που είναι ντυμένη. Όμως οι τεχνικές είναι όλο και πιο εξελιγμένες, φτιάχνουν ειδικέ στολές για τη μεταφορά παράνομων ε, προϊόντων και ε, ο σκοπός να αποφύγουν τον αντοπισμό με το να φαίνεται φυσιολογική η κορμοστασιά τους και η ενδυμασία τους ένα ζωντανό ε, τυγράκι που είχε ναρκωθεί και είχε συσκευαστεί μαζί με ψεύτικα λούτρινα τυγράκια. Εδώ βλέπετε μία μεταφορά ελεφαντοστού, ελεφαντόδοτου. Η ποιότητα και η έλλειψη κρυψίματος εδώ, ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να κρυφτεί, σημαίνει ότι υπάρχει συνενοχή μέσα στο σύστημα. Επομένως ε, πρέπει να εντοπίσουμε και να ε, αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ας δούμε την αντίχνευση και χαίρομαι διότι αναφέρθηκαν οι ακτίνες Χ. Ποια είναι η πρόκληση, η ιεράρχηση, το να δοθεί προτεραιότητα στο ένα ή στο άλλο. Η τελωνία κυρίως ενδιαφέρονται για παραποιημένα προϊόντα ή για προϊόντα που δημιουργούν κίνδυνο ασφάλειας. Ενώ η άγρια πανίδα ε, δεν είναι ούτε, δεν έχει ούτε κίνδυνο ασφάλειας απαραίτητα ή πάντοτε, ούτε είναι παραποιημένη. Ε, μπορεί εδώ ε, ό,τι φαίνεται πορτοκαλί να ε, έχει κόκκινη σημαία γιατί φαίνεται ότι είναι ζώσα ζωή. Δεξιά όμως είναι πράγματα πράσινα και μπλε δηλαδή που δεν εγείρουν ανησυχίες. Ενώ ουσιαστικά όταν ανοίξαμε είδαμε ότι είναι ελεφαντόδοτο. Έχουμε κάποιες περιπτωσιολογικές μελέτες και τις δείχνουμε στις εταιρείες για να τους δείξουμε πώς χρησιμοποιούν τα συστήματά τους και τι κάνει ο κόσμος για να παρακάμψει τις πολιτικές της εταιρικές έτσι ώστε ε, να μεταφέρει αυτό που θέλει. Σε αυτές τις περιπτώσεις Δώσαμε παραδείγματα πολλαπλών διελεύσεων και διαδρομών που χρησιμοποιούνται για να αποφύγει κανεί τον εντοπισμό. Μία φορά περνάει από το ένα μέρο στην άλλη από το άλλο. Υπάρχουν λιμένε με λιγότερη ασφάλεια που είναι γνωστό αυτό. Εξετάζουμε περιπτώσεις χαμένων αποσκευών όπου μετά έρχεται ε, κάποιος και παίρνει τη βαλίτσα αργότερα. Έχουμε, εξετάζουμε πακέτα που ε, περιγράφονται ως κάτι που δεν είναι αλλά και συσκευασίες που κυκλοφορούν πάνε μπρος πίσω μέχρι ότου βρεθεί ε, μια, ε, βρεθεί μια στιγμή όπου η ασφάλεια είναι ελληματική. Για παράδειγμα, μια ε, βαλίτσα παραδόθηκε όταν τα ειδικά σκυλιά τα ανείχνευσης δεν βρίσκονταν στο αεροδρόμιο και ήταν γνωστό αυτό. Τότε μόνο ζητήθηκε δηλαδή για να την παραλάβει ο ενδιαφερόμενος. Όλα αυτά τα έχουμε δείξει επανειλημμένως στους πελάτες και υπάρχουν και στα αεροδρόμια. Προσπαθούμε όμως να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση και μέσα στο ε, ε, στον ιδιωτικό τομέα. Δίνουμε υλικό, ε, δίνουμε κατάρτιση. Υπάρχει ζήτηση για όλο και περισσότερες πληροφορίες είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς πώς θα επικοινωνεί με τις τελωνιακές αρχές. Πολύ συχνά μας λένε ότι παρόλο που οι ιδιωτικές αρχές ήξεραν με ποιον να έρθουν σε επικοινωνία στον ιδιωτικό τομέα, οι ιδιωτικές εταιρείες μας λένε ότι δεν ήξεραν με ποιον να έρθουν σε επικοινωνία από πλευράς διοκτικών αρχών και αυτό δεν ισχύει. Είναι γνωστή η τηλεφωνική αριθμή. Επομένως, Πρέπει να πω ότι ο ιδιωτικό τομέα δεν είναι ειδικό στην ταυτοποίηση των ειδών και ούτε θα έπρεπε να είναι, αλλά θα έπρεπε να ξέρει ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσει ώστε να πάρει βοήθεια. Πρέπει να δούμε και τους κινδύνους που υπάρχει η μεταφορά της άγριας πανίδας, όχι μόνο από την πλευρά των ζώων, αλλά και από την πλευρά της υγείας και ε, της πολιτικής υγείας. Το να μεταφέρει κανείς άγρια πανίδα πάνω στο σώμα του ή να το βάλει σε μια βαλίτσα δεν, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Και είναι ένας κίνδυνος υγείας, γιατί μπορεί να μεταδοθούν νοσήματα, ανθρωποζωονόση και ε, υπάρχουν ζώα που είναι επικίνδυνα, δηλητηριώδη και αυτό γύρουν ζητήματα ασφαλείας και δημόσιας υγείας. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν είναι ότι υπάρχει επιθυμία να μοιράζονται περισσότερες πληροφορίες ιδιωτικό τομέα με τις διοκτικές αρχές και στη συνέχεια να αναλαμβάνεται δράση. Το έγκλημα, το λαθρεμπόριο άγρια πανίδα θα πρέπει να αναβαθμιστεί, δηλαδή η αξιολόγησή του να θεωρηθεί ότι είναι ένα από τα σοβαρά διεθνή εγκλήματα για να ε, Και ο ο Φαντουίν ο οποίος είναι συντονιστής ε, ασφάλειας της Ιντερπολ και επομένως εστιάζει κατευθείαν στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χρειάστηκε να, προβα... να προφέρετε τρία Ολλανδικά ονόματα, Ντόιν λέγουμε. Είναι μεγάλη πράγματι αυτή η πρόκληση. Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας και μπορώ να λάβω το λόγο ενώπιον της Επιτροπής του Ευρωβουλίου ε, εξ ονόματος της Ιντερπολ. Δυστυχώς δεν έχω μια εικόνα η οποία συμπληρώνει αυτή της ε, Μισελ. Όταν δούλευα στην αστυνομία του Ρότερνταμ, πιάσαμε ένα λαθρέμορο, ο οποίος είχε στα εσώρουχά του οδικά πτηνά. Είχε δέκα πουλιά λοιπόν που τα είχε στα εσώρουχά του. Και όταν τον ρωτήσαμε στη συνέχεια, γιατί το κάνατε αυτό, γιατί βάλατε τέσσερα δέκα πουλιά στα ρούχα σας. Το ξέραμε ότι μετέφερε ναρκωτικά συνήθως. Είπε, κύριε Φοντάιν, αυτό βγάζω πιο πολλά λεφτά με αυτό το, με αυτό το λαθρεμπόριο. Πουλούνται για 6.000 ευρώ το ένα τα πουλιά αυτά. Και το μεγαλύτερο πρόστιμο που θα μπορούσατε να βάλετε είναι 500 ευρώ και ενδεχομένω θα μου δώσετε πίσω και τα οδικά πουλιά. Επομένως αυτά τα υψηλά κέρδη και τα χαμηλά πρόστιμα οδηγούν στο λαθρεμπόριο αυτό. Ο στόχος μας είναι λοιπόν να πείσουμε τις χώρες όλου του κόσμου να αντιμετωπίσουν το σοβαρό έγκλημα για τα θέματα αυτά. Ένα από αυτά τα σοβαρά εγκλήματα είναι εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος. Από το 2014, σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβάλλοντος του ΟΗΕ, έχει αυξηθεί σημαντικά το το έγκλημα κατά του περιβάλλοντος κατά 26%. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το πόσα χρήματα εμπλέκονται, ποιος είναι ο σωστός ορισμός για το έγκλημα αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε κάτι μεταξύ 91 μέχρι 250 ε, εκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια το χρόνο σε κέρδος. Είναι περίπου διπλάσιο το, από το συνολικό ποσό που χρησιμοποιείται για αναπτυξιακή βοήθεια σε πολλές χώρες. Το έγκλημα για το, κατά του περιβάλλοντο, είναι οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια που γίνεται από εγκληματικές οργανώσεις για να παράγει κέρδη, τα οποία όμως οδηγούν σε μεγάλη ζημιά προς το περιβάλλον. Όχι μονάχα είναι μια απειλή προς το περιβάλλον αυτό το έγκλημα, αλλά θίγει και τα έσοδα των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων και μειώνει τη δυνατότητα αηφόρου ανάπτυξης και είναι και εμπόδιο στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί από αυτού που ασχολούνται με το έγκλημα κατά του περιβάλλοντο, <clears throat> προέρχονται από άλλους εγκληματικού τομεί και έχουν διευρύνει τις δραστηριότητε τους και στο περιβάλλον και ασκείται από προηγούμενα δίκτυα εγκληματικού χαρακτήρα λόγω του, της κερδοφορία του συνδέεται με το κυβερνό έγκλημα, την λαθεμπορία ναρκωτικών, τα χρηματοπιστωτικά εγκλήματα, τη διαφθορά υπάρχουν και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία. Από την πλευρά της Europol έχουμε δυσκολίες να καταδείξουμε ότι συνδέεται με την τρομοκρατία αυτό το έγκλημα, αλλά είναι σαφώς, σαφές ότι υπάρχουν τέτοιες πτυχές. Είναι ιδιαίτερα λοιπόν σημαντικά αυτά τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος και επιπλέον ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα και την έκταση αυτών των εγκλημάτων είναι απαραίτητο να τα αντιμετωπίσουμε αυτό προ όφελο των κρατών μελών. Το 2015 σε ερωτηματολόγιο η Europol έχουμε ένα γραφείο σε κάθε χώρα για να ασχοληθεί με τα θέματα αυτών των προτεραιότητων για το περιβαλλοντικό έγκλημα. Η απάντηση, η απάντηση δείξα ότι είναι εθνική προτεραιότητα για 87% από τις χώρες που απάντησαν και πάνω από 60% απήντησαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο. Λόγω λοιπόν της δέσμευσής μας να υποστηρίξουμε τις <clears throat> χώρες μέλη. Πρέπει να, να αντιμετωπίσουμε και το θέμα αυτό. Ο αγώνα κατά το εγκλήματο του περιβάλλοντο όμω δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα. Πρέπει να υπάρχει μια παγκόσμια και συνεργατική προσπάθεια. Και εγώ προσωπικά ως αστυνομικός έχουμε, όταν έχουμε μια περίπτωση αυτού του είδους προφανώς εμπλέκονται πολλοί υπαλληδιοκτικού διοκτικού χαρακτήρα, πολλές φορέ δεν συνεργαζόμαστε και στα εγκλήματα κάτω του περιβάλλοντος επειδή υπάρχει πολυπληθώρα αρμοδίων είναι υποχρεωτική η συνεργασία. Χρειάζεται να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία των αστυνομικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο υπό την αιγύδα τη Interpol και με τη βοήθεια των Εθνών και του ιδιωτικού τομέα. Χαιρόμαστε λοιπόν που η Interpol υπέγραψε μια συμφωνία με το Αμερικανικό με το πρόγραμμα του ΟΗΕ για την εφαρμογή κανόνων δικαίου στο περιβάλλον. Αυτή η συμφωνία ενισχύει και τους θεσμούς που έχει ήδη η Europol με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και θα επιτρέψει την ανάπτυξη προγραμμάτων υψηλού επίπεδου που θα αντιμετωπίσουν το έγκλημα και επίσης θα βοηθήσει την πρόσβαση σε πλατφόρμες όπως το Ταμείο για την ε, προστασία του περιβάλλοντος. Σας λέω και πάλι ότι είναι απαραίτητες οι συνεργασίες για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Το 2014, όπως είπα, ο συναδελφός μου, η Interpol και άλλες τέσσερις διακυβερνητικές οργανώσεις άρχισαν να εργάζονται από κοινού για ένα διεθνές consortium, το IQIC, για την αντιμετώπιση του ε, λαθεμπορίου αγριων Με μπερδεύει και εμένα, επειδή δεν είναι η μυητική μου γλώσσα τα αγγλικά, το ΑΕΚΟΙΚ όμως συνδέει πέντε οργανώσεις, τον Διεθνή Οργανισμό Τελωνίων, την, ε, τη, το Γραφείο των ΗΠΑ για το έγκλημα και το, τα ναρκωτικά, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους φορείς. Για να μπορέσουμε λοιπόν να λειτουργήσουμε χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία και σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τα εγκλήματα στο τομέα του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα για το 2017-2020 που έχει παρουσιαστεί στη διεθνή κοινότητα των χορηγών για να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε τα αποτελέσματα τα οποία επετέθησαν μέχρι σήμερα. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητε <clears throat> και δεν μπορούμε να τις παρουσιάσουμε δυστυχώς όλες, αυτή τη στιγμή χρηματοδοτεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φέρνουν έτσι την συνεισφορά του όλοι οι οργανισμοί που συνεργάζονται για τα θέματα αυτά. Και αυτή η υποστήριξη που προέρχεται από αυτού του τομεί δίδεται σε όλη την αλυσίδα εφαρμογής για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Ξεκινήσαμε από συλλογέ δεδομένων και φτάσαμε σε επίπεδο εισαγγελιών και δικαστικών διώξεων. Ένα από τα προϊόντα είναι η επανεξέταση, αν θέλετε, η αξιολόγηση του πού βρισκόμαστε σε σχέση με ρυθμίσεις που έχουν ισχύσει στο παρελθόν. Θέλουμε λοιπόν ένα νέο πλαίσιο για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Και εμείς και άλλοι εταίροι προσπαθούμε να δούμε πώς θα εξαλειφθεί το πρόγραμμα αυτό μέχρι το 2020. Ε, επίσης θα συζητηθεί και το Νοέμβριο από την ε, σειρά των δωρητριών χωρών. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλές οργανώσεις, σε task force που έχουν σαν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε εμείς να καταστήσουμε προσβάσιμο για το κοινό και τους εργαζομένους στις μεταφορές να δίδουν πληροφορίες για ποινικά κολάσιμες δραστηριότητες. Είναι πολύ δύσκολο να βρίσκει κανείς τέτοιου είδους στοιχεία και γι' αυτό προσπαθούμε με ένα διακριτικό τρόπο να συνεισφέρουμε κι εμείς. Σε όλο τον κόσμο ζητάμε πολλά μένα από τις ε, επιχειρήσεις, αλλά θέλουμε τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν να βοηθήσουν σε επίπεδο αηφορίας και ανάπτυξης. Εμείς ε, επίσης έχουμε κάποιους στόχους για την καταπολέμηση των ε, ποινικών παραβιάσεων γενικά στον τομέα της παραγωγής προϊόντων σε σχέση με την παράνομη δασοκομική δραστηριότητα εμείς θέλουμε να σταματήσουμε τις τάσεις οι οποίες οδηγούν στην μείωση των εκτάσεων με δάση και στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική και την Ασία. Πολλές φορές εισάγονται σε ορισμένες χώρες ξυλία, η οποία, η προϊόντα ξυλίας όπως χαρτί και ε, άλλες μορφές, αλλά πρόκειται για επεξεργασμένα προϊόντα που προέρχονται όχι από τη χώρα εξαγωγής, από χώρες διαφορετικές. Έχουμε διακόψει τη λειτουργία πολλών ε, εγκληματικών δικτύων, τα οποία όμως εξακολουθούν να είναι στον τομέα σαν παράδειγμα των μεταφορών δραστήριες. Είδαμε να αναμειγνύεται ο άνθρακας σαν παράδειγμα με το ελεφαντόδοντο. Επίσης έχουμε ασχοληθεί και με τις πληροφορίες που μας έχουν δώσει διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να αποκτήσουμε πληροφορίες και να ενημερώσουμε τις κατασταλτικές αρχές. Επίσης ε, προσπαθούμε και με το πρόγραμμα Infotera έχουμε επίσης ε, ε, διακόψει και εγκληματικά δίκτυα και στις χώρες προέλευσης και στις χώρες εμπορίας. Είναι πολλές δραστηριότητες βέβαια δύσκολο να ανοιχνευθούν από τις υπηρεσίες της αρμόδιες, αλλά προσπαθούμε να πείσουμε τις αρχές καταστολής ότι ναι μεν υπάρχουν άλλες προτεραιότητες όπως η καταπολέμηση της εμπορίας των όπλων, η τρομοκρατία κτλ. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια πρόκληση ενδιαφέροντος και για τα θέματα που μας αφορούν. Ε, πρέπει να αυξήσουμε και τις δυνατότητες παρέμβασης Υπάρχει σε επίπεδο WCO ε, η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον περισσότερο. Θα τελειώσω αγαπητοί συνάδελφοι λέγοντας ότι η Interpol είναι μη πολιτική οργάνωση η οποία εμπλέκεται σε διαδικασίες δίωξης κάποιων δραστηριοτήτων με ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση. Απαιτείται λοιπόν μια αποτελεσματική μορφή ανταλλαγής πληροφοριών και συνδυασμού των προσπαθειών, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να είναι πιο αποτελεσματικές. Αυτό θα βοηθήσει και με την, θα βοηθηθεί και με την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα. Η Interpol είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην παγκόσμια κοινότητα για την βελτίωση των συνθήκων ασφαλείας που άπτονται του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ. Στη Γερμανία έχουμε το DUN που το ίδιο προφέρεται, δεν δυσκολεύτηκα και πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Έμα. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Νομίζω ότι μας εμπνέει πραγματικά να ακούμε τη δράση σας, ειδικότερα εσάς κυρία, κύριε Κάουτσμαν. Είδαμε πόσο ο ιδιωτικό τομέα δήλωσε παρόν σε αυτόν τον αγώνα μετά τη δήλωση του Buckingham Palace. Όμως οι βελτιώσεις των Φιλιππινών πώς μπορούν να υιοθετηθούν ως πολιτικοί. Και απευθύνω το ερώτημα σε όλους σας. Τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα κάνει τη διαφορά και κύριε Ντούιν από την Ίντερπολ. Ποιο είναι αυτό το ένα πράγμα που μπορούμε εμείς εδώ να κάνουμε για να ε, ε, ε, ε κάνουμε τη διαφορά στην καθημερινότητα των διοκτικών αρχών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές γιατί με τον τρόπο με τον οποίο έχουν παρουσιάσει την κατάσταση είναι σαφές το ποια είναι η πραγματικότητα και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει η κοινή γνώμη όπως θα έπρεπε να το γνωρίζει. Θα ήθελα να σταθώ στο εξή το οποίο αναφέρατε όλοι, ότι στη διαδικασία μεταφοράς αυτών των αγαθών στα τελωνία να αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, διαφθοράς. Και επανέρχομαι στο πρόβλημα αυτό το οποίο αναφέρθηκε, ότι πολλές φορές έχουμε ζώα τα οποία είναι νεκρά, έχουν ήδη σκοτωθεί όταν μεταφέρονται. Πρέπει λοιπόν το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί στην πηγή, να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών και των ΜΚΟ για να εμποδιστεί η σύλληψη αγριών ζώων οι δασοφύλακες, οι, οι rangers οι οποίοι είναι στα, στους χώρους όπου ζουν τα άγρια ζώα, αυτοί θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη υποστήριξη και να έχουν και τον κατάλληλο εξοπλισμό για να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν την αξία που έχει η φύση και η προστασία της και αυτό σημαίνει ότι πρέπει και ο τουρισμός, είτε πρόκειται για σαφάρι, είτε πρόκειται για φωτοσαφάρι, να χρησιμοποιηθούν τα έσοδά του για να προστατευτεί η φύση και είναι απαραίτητο να γίνουν αυτές οι ενέργειες γιατί χάνουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος ε, και, στις, ε, και στην ε, ε και στην κατανάλωση κρέατος από άγρια ζώα και αυτό είναι κάτι το μπούσμι το οποίο δεν πρέπει να το παραμελήσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Δίνω του εμπειρογνώμου και πάλι τον λόγο για να απαντήσουν εάν το επιθυμούν. Οι καλεσμένοι μας από το Βιετνάμ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για τα σχόλια που αναφέρθηκαν, πράγματι πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα για να βελτιώσουμε την συνειδητοποίηση της κοινή γνώμης σε σχέση με το πρόβλημα και την ανάγκη προστασίας των αγρίων ειδών. Ένα από τα εργαλεία για να υπάρχει αυτή η προστασία είναι να του ενθαρρύνουμε να αναφέρουν παραβιάσια τα θέματα αυτά. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή στην οποία μπορούν να καταγγείλουν οι πολίτες. Πρέπει φυσικά όμω να, να έχουμε και μια παιδαγωγική δράση εναντίον των ανθρώπων και να του εξηγήσουμε την ανάγκη να προστατεύσουν την ε, άγρια ζωή. Αυτό είναι μια μακροχρόνια επένδυση. Γι' αυτό ένα τμήμα των προσπαθειών μας είναι να αποθαρρύνουμε την κατανάλωση κρέατος από άγρια ζώα επειδή είναι αργά όταν έχουν ήδη σκοτωθεί τα ζώα, πρέπει να υπάρξει αποτελεσματική πολιτική για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι απάντησε στο ερώτημα. Ευχαριστώ, λέει και ο Δύο ερωτήματα, σε δύο ερωτήματα θέλω να απαντήσω για το μοίρασμα των δεδομένων. Ο συνάδελφος από την Interpol το είπε ότι μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες μεταξύ ΠΟΕ και Interpol και νομίζω ότι πολλές τελωνιακές διοικήσεις ακολουθούν αυτό το δρόμο. Είναι πιθανό λοιπόν, είναι εφικτό και θα ήταν εξαιρετικά ισχυρό ως εργαλείο που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Τώρα, οι φίλοι μου στην Τανζανία και στην Κένια είναι πεπισμένοι ότι η παλαιότερη γενιά δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει διαφθορά μεγάλη στην υποσαχάρια Αφρική και θα είναι δύσκολο να αντιστραφεί το κλίμα. Ε, θεωρούν ότι υπάρχει μια ευκαιρία με τα παιδιά. με τους νέους ανθρώπους και γι' αυτό οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ασχολούνται κυρίως, έχουν κυρίως δράση μέσα στα σχολεία ε, για να καταρτήσουν τη νέα γενιά και νομίζω ότι αυτό είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Όμουεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως προς την εκπαίδευση και τις εκστρατείες συνειδητοποίησης και ενημέρωσης, είναι πολύ κρίσιμο ζήτημα, πολύ σημαντικό, συμφωνώ. Ε, είναι ένα ζήτημα που επιτυχάνεται σε βάθος χρόνου. Πάρα πολλές επενδύσεις γίνονται σε τέτοιου είδους εκστρατείες, προσπαθώντας να αλλάξουν τα στερότυπα και οι προκαταλήψεις προσπαθώντας να αλλάξουν τους λόγους για τους οποίους να θέλει κανείς να αγοράσει ένα προϊόν της άγριας πανίδας. Ουσιαστικά αναγνωρίζουμε ότι δεν θα λυθεί το πρόβλημα με όλες αυτές τις εκστρατείες ενημέρωσης. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα εξαιρετικά καλά οργανωμένη και πρέπει να παταχθεί σε πολλαπλά επίπεδα και γι' αυτό λαμβάνει δράση ο ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να επιβληθεί ο νόμος, πρέπει να υπάρχει δίωξη και πρέπει να είναι συνδυασμένη προσπάθεια και σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε εκπαίδευση και συνειδητοποίηση και ούτω καθεξής. Παρακαλώ κύριε Φοντόιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με ιντρικάρει αυτό το ερώτημα ποιο είναι το μόνο πράγμα, το ένα πράγμα που να αφαιρώσουμε πόρους εκεί για να αλλάξουμε την κατάσταση στη θέμελα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν έχω τέτοια απάντηση. Νομίζω ότι ασχολείται με αυτό το θέμα η διάσκεψη των μερών ε, στο Λονδίνο με τη δήλωση του Κασάνε και στο Ανόη θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό αργότερα. Ε, για να αποσταματήσει η λαθροθυρία που σχετίζεται ε, αυτό και με αυτό που είπε ο κύριος Όμπερμαερ και έχει απόλυτο δίκιο. Από πλευράς Ιντερπολ είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τις διοκτικές αρχές και κυρίως το ερευνητικό τους έργο. Τώρα, αν θέλουμε αυτό να το βελτιώσουμε, ε, τότε να δίνονται οι πόροι σε μια βιώσιμη στήριξη και ενίσχυση των διοκτικών αρχών και ενθάρρυνση, να δίνονται πορεί στην ενθάρρυνση συνεργασίας αστυνομικών τελωνιακών, αστυνομικών ε, δασικών ε, υπαλλήλων. Να υπάρχουν κοινέ ε, ομάδες, μικτές ομάδες που να δραστηριοποιηθούν επί τόπου. Και ίσως αυτό θα διευκολύνει και την ανταλλαγή πληροφοριών μακροπρόθεσμη βάση. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ολοκληρώνεται νομίζω η συζήτησή μας για το θέμα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τους παρισταμένους, τους παρόντες, τους εμπειρογνώμονες, κυρίως την εκπρόσωπο, ε, την προσκεκλημένη μας από το Βιετνάμ, η οποία διάνυσε τόσο μεγάλη απόσταση για να είναι εδώ μαζί μας. Χαίρομαι διότι έχουμε συζητήσει εκτεταμένα τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ε, με το Βιετνάμ και η παρέμβασή σας ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια σημαντική αγορά ε, και άρα προορισμό ε, των προϊόντων λαθρεμπορίου άγριας πανίδας. Ο εκπρόσωπος της Ιντερπόλ σας είπε ότι αυξάνεται το λαθρεμπόριο άγριας πανίδας και δεν είναι καθόλου θετικό αυτό το μήνυμα το οποίο ε, λαμβάνουμε σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε το παν για να αλλάξουμε το τοπίο. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα αυτό. Σήμερα έμαθα ότι η πολιτική μας πρέπει να... Το σημαντικότερο είναι να είναι συνεκτική, να έχει συνέπεια. Και είναι κάτι πολύ βασικό και στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουμε και στην εφαρμογή όλων αυτών των συμφωνιών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, με τις τρίτες χώρες και ε, στις εταιρικές σχέσεις μεταξύ ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και πρέπει να κάνουμε το παν για να ενημερώνουμε το κοινό αλλά να ενημερώνουμε και τον μηχανισμό, τον διοικητικό μηχανισμό. Είναι τεράστιες οι προκλήσεις στα σύνορα, στους λιμένες της Ευρώπης. Πρέπει να δώσουμε στα τελωνία περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ικανότητες για να μπορέσουν να ελέγξουν και να ε, συντονίσουν τις προσπάθειές τους καλύτερα, έτσι ώστε όλοι να κάνουμε ένα βήμα που είναι τόσο απαραίτητο σε αυτή την προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου άγριας πανίδας. Την έκθεση για το θέμα αυτό θα την εξετάσουμε στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, γνωρίζει το θέμα και το έχει υπόψη της και θα το έχει υπόψη της και για τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες που θα εξετάσει έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ό,τι παλαιότερα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επομένως, προχωρούμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης, εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Να δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή μας, ε, Εμμανουέλ Μορέλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί δεν θέλω να κουράσω τους συναδέλφους. Νομίζω ότι συμμεριζόμαστε όλοι στη διάγνωση που έχουμε ε, κάνει. Η Ευρώπη έχει ζωτική ανάγκη επενδύσεις, επενδύσεις ιδιωτικές και δημόσιες, το σχέδιο Juncker όπως έχει αποκληθεί και σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε η Επιτροπή μας να συντάξει ένα σχέδιο γνωμοδότησης για τη νέα ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος υπογράμμισε τη βούλεσή του να δώσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων ένα εξωτερικό σκέλος, μια εξωτερική διάσταση τάση για να υπάρχουν αναπτυξιακές επενδύσεις στις χώρες γειτονίας και στις τρίτες χώρες. Σας προτείνω λοιπόν να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα ε, υπό τον όρο όμως ότι συγκεκριμένε αρχές θα ε, τηρούνται. Σίγουρα ε, είναι ένας καμβάς αυτό ε, το κείμενο να σας πω καταρχάς ότι είναι ένα εργαλείο στη διάθεσή μας, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτεί επιπρόσθετα project, δηλαδή έργα που ε, ε, έχουν κίνδυνο, έργα που είναι καινοτόμα στην ενεργειακή μετάβαση, στη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, ε, έργα δηλαδή που δεν θα υπήρχαν χωρίς την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Από εκεί και πέρα για να είναι αποτελεσματικός ο μηχανισμός θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δώσουν ρευσότητα υπό τη μορφή εγγυήσεων. Δέκα κράτη-μέλη το έχουν κάνει, αλλά θα πρέπει αυτό να ισχύσει και για τις τρίτες χώρες και κυρίως την Κίνα. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, θέλω να γραφτεί ξεκάθαρα ότι η Κίνα, αν θελήσει να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση τέτοιου είδου έργων, δεν θα πρέπει να περιμένει κανένα αντάλλαγμα ή καμία κανένα αντιστάθμισμα. Θα πρέπει να έχει επιλέξει μόνη τη να επενδύσει για του δικού τη λόγου. Θέλω αυτό να αναγραφεί ξεκάθαρα. Ε, από ό,τι ε, ε, γνωρίζω από τη Γαλλία και νομίζω ότι ισχύει και στην Ιταλία ότι προβλέπει το σχέδιο Juncker για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι θετικό. Θα πρέπει να τις βοηθήσουμε στη διεθνοποίησή τους γιατί αυτές είναι που δημιουργούν και το μεγαλύτερο και περισσότερο πλούτο και προτείνω να διευρύνουμε την σχετική πλατφόρμα και να της δώσουμε τη δυνατότητα ε, να, μεταξύ των ε, καθηκόντων της να είναι και η βοήθεια προς τις εξαγωγές. Είχε ανακοινωθεί ένα επενδυτικό σχέδιο για τις χώρες της Αφρικής ε, και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας μεταξύ 44 και 88 δις ευρώ. Είναι εξαιρετικά φιλόδοξο το σχέδιο αυτό. Προτείνω λοιπόν οι επενδύσεις που γίνονται ε, βάσει σχεδίου Juncker να προστίθεται στις υφιστάμενες επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή της Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. Δηλαδή να έχουμε την αρχή της προσθετικότητας. Και παρόλο που πιστεύω ότι συμφωνείτε ούτως ή άλλως, να πω ότι ε, σκοπός είναι και πρέπει να αναγραφεί ότι ε, δεν είναι ο σκοπός να κερδοσκοπήσουμε στην πλάτη των Αφρικανών, αντισέτως να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες, ε, ειδικότερα σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές όπου είμαστε μάρτυρας, μάρτυρες όλοι της συλλογική εξόδου των λαών αυτών από τον τόπο τους. Σας ευχαριστώ και ελπίζω για τη στήριξή σας για αυτή την έκθεση η οποία είναι πολύ σύντομη πράγματι και παρόλο που είναι μόνο σχέδιο γνωμοδότησης, πιστεύω ότι είναι σημαντικό ε, να επενδύσουμε περισσότερο ε, στο μέλλον για να το προετοιμάσουμε και καλύτερα άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρος. Ο... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ρούας, ότι θέλω να εξάρω το έργο του εισηγητή Νομίζω ότι το Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων θα πρέπει να κατευθυνθεί προς την βιομηχανία που είναι μια βασική πηγή πλούτου σε μια ε, οικονομία η οποία είναι ανταγωνιστική. Θέλω να προσθέσω όμως ότι, ότι μπορεί να βοηθήσει και την ε, δημόσια δίκηση και την αποτελεσματική διακυβέρνηση. Και επίσης είναι σημαντικό όπως λέγεται και στην έκθεση να λάβω υπόψη ότι η συμμετοχή της Κίνας σε αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης δεν πρέπει να οδηγήσει σε αντισταθμίσματα, όπως παραγωγή χάρη η χορήγηση στη χώρα αυτή του χαρακτήρα χώρας με οικονομία της αγοράς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι θα πλητανεύουν οι κανόνες του ΠΟΕ στο διεθνές εμπόριο, Πρέπει επίση να υπογραμμίσω τη σημασία των προτάσεων που έχει υποβάλει ο πρόεδρο Γιούγκερ στην ομιλία του για την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ανάγκη, τονίζοντα να υπάρχει και μια εξωτερική πτυχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει και σε εσωτερικό επίπεδο και σε εξωτερικό επίπεδο. Επίση, ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του Ταμείου αυτού, η διαδικασία επιλογή των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι διάφανη και αυστηρή <clears throat> και όχι ε, προς ε, το συμφέρον ορισμένων επιχειρήσεων, θα πρέπει να ευνοηθεί η πλατφόρμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εξωτερικό εμπόριο, που είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι το 98% του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού ιστού και επομένως η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Γι' αυτό το λόγο το σχέδιο επενδύσεων και το σχέδιο Juncker θα πρέπει κατά την άποψή μου να εστιαστεί στην διεθνοποίηση, την υποστήριξη των εξαγωγών και μια καλύτερη ομοιογενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική πρέπει το Ταμείο αυτό να προωθήσει καλύτερη ισορροπία σε γεωγραφικό επίπεδο και εξασφάλιση ομοιογένεια σε ε, γεωγραφικό επίπεδο της οικονομίας των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τις τρίτες χώρες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την πρόθεση των στόχων του Ταμείου σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να λειτουργήσει το Ταμείο αυτό σε προσθετικότητα και συμπληρωματικότητα με, τους άλλους, με τα άλλα ταμεία διαδοτικού χαρακτήρα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις μεταναστεύσεις και τις βαθιές αιτίες τους, γιατί αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, είναι απαραίτητο ένας από τους κύριους στόχους του Ταμείου είναι να αντιμετωπίσει τις μεταναστεύσεις επί τη βάση των αρχών της ανάπτυξης και της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υποστηρίξουμε και διαμεθοριακά σχέδια τα οποία δίδουν προσθεμένη αξία στον επιχειρηματικό τομέα και τελευταίο σημείο, το οποίο όμω δεν είναι και το ίστατο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρακολουθιστεί η εφαρμογή αυτού του Ταμείου και να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για το μέλλον. Αυτά είναι τα σημεία που ήθελα να παρουσιάσω, κύριε Πρόεδρε, και θα παρουσιάσω φυσικά και ορισμένε τροπολογίε προ αυτή τη γνωμοδότηση που θα αντανακλούν αυτά που σα είπα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λούνς για τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά. Εμείς θα υποστηρίξουμε τις βασικές αρχές της πρότασης. Υποστηρίζουμε κυρίως την παράγραφο 3 για την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων. Θεωρούμε ότι είναι μια προτεραιότητα και απαιτείται να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Hub ενίσχυση των μικρομεσαίων. Εγώ ήμουν εισηγητής για το θέμα αυτό στην ΕΚΟΝ, το είχαμε συζητήσει, τώρα είναι πάλι υποσυζήτηση. Νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός. Δευτέρον, θα συμφωνήσουμε επίσης και με το εξωτερικό στοιχείο του Ταμείου αυτού, το οποίο είναι υποσυζήτηση και αυτό είναι συμβατό με τις πολιτικές μας στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης και η αναπτυξιακή βοήθεια είναι ε, βασική πηγή χρηματοδότησης για πολλές χώρες και θα πρέπει να εμπλακεί εδώ και ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας γίνεται σταδιακά συμπλήρωμα των κυβερνητικών οργανώσεων και του δημοσίου, ένας εταίρος πλήρης πλέον που συμμετέχει στον καθορισμό των στρατηγικών μας, ε, και που ε, ενισχύει την αναπτυξιακή βοήθεια και τις δανειοδοτικές δραστηριότητες. Ανοίγει λοιπόν νέες δυνατότητες για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τελευταίο στοιχείο, αυτό το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην παράγραφο εδώ είναι η σημασία των επενδύσεων αυτών στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσθεθεί σε αυτά τα οποία προτείνεται. Και γι' αυτό θα κατατεθεί μια τροπολογία. Ευχαριστώ πάντως είναι μια καλή στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική πλέον. Και η Σκά Κέλλερ αντικαθιστώντας τον Ζαντό. Εγώ είμαι η σκιώδης εισηγήτρια, αλλά εντάξει. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Είναι θετική η πρότασή σας. Αυτό το οποίο μας ικανοποιεί είναι αυτό το οποίο λέτε ότι οι δραστηριότητες του ΕΦΣΥ, του Στρατηγικού Ταμείου, θα πρέπει να είναι συμβατές με τις δραστηριότητες της Ένωσης στον εξωτερικό τομέα και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για την καταπολέμηση των αιτιών που οδηγούν στη μετανάστευση. Εγώ δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ΕΦΣΥ για να κάνουμε συμφωνίες για επανεντάξεις, για επανεισδοχές μάλλον αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τις πραγματικές αιτίες της φτώχειας, της έλλειψης προοπτικής και της μετανάστευσης τελικά. Δεν πρέπει λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε σαν μοχλό για συμφωνίες επανεισδοχής. Θα συμφωνήσω με την πρόταση του εισηγητή ότι οι μελλοντικέ δραστηριότητες του Στρατηγικού Ταμείου θα πρέπει να είναι συμβατές με την αρχή της προσθετικότητας σε σχέση με αυτά που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και να καλυφθούν επίσης και προγράμματα μικρότερης κλίμακας και με υψηλότερους κινδύνους. Υπάρχουν δύο τομείς στους οποίους δεν είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Το ένα είναι η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διευκρινίσει ιδιαίτερα διότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι ιδιαίτερα δραστήριες και παρούσες στις επενδυτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ασία. Έχουμε επιφυλάξει γι' αυτό και επίσης για τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων. Αν θέλουμε να το πούμε αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε πως κάτι τέτοιο μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί έτσι όπως λειτουργεί το ΕΦΣΥ, στην ουσία οδηγεί στο να κατανεμηθούν πολύ ψηλά ποσά σε ορισμένους χώρους που δεν καλύπτουν τις μικρομεσαίες. Γι' αυτό λοιπόν εδώ έχουμε ένα ερωτηματικό. Ο κύριος Τάκουλας. Κυρία Ντεσάνες δεν μπορεί να είναι εδώ παρούσα σήμερα, γι' αυτό θα ήθελα να την αντικαταστήσω και θέλω να ευχαριστήσω εξ ονοματός της τον εισηγητή που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων έχει δημιουργηθεί πριν από ένα χρόνο και παραπάνω. Τα αποτελέσματά του μέχρι στιγμή συνολικά μπορούν να θεωρηθούν πολύ ικανοποιητικά. Το 1 τρίτο περίπου των 315 δισεκατομμύρων που προβλεπόταν έχουν κινητοποιηθεί για επενδύσεις. 62 σχέδια έχουν και ιδιωτικές επενδύσει ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση του ΕΦΣΥ θα ήθελα να αναφερθώ στου εξή τομεί. Πρώτα απ' όλα τα ταμεία του EFSI θα πρέπει να εξυπηρετήσουν ευρωπαϊκά συμφέροντα και να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Δεύτερον, θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και να κάνουμε μια διαφοροποίηση των πηγών κεφαλαίων. Δεν πρέπει να εξαρτώμεθα από την Κίνα. Επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε την διεθνοποίηση της δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι κέρια σημασία. Τέταρτον, θα πρέπει να αναπτύξουμε μια εξωτερική διάσταση για το ΕΦΣΥ με στοχοθεσία και συνεκτικούς στόχους οι οποίοι να παραμείνουν να συνάδουν με τη λειτουργία του ΕΦΣΙ στην Ευρώπη. Και τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλει στην βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος στην εσωτερική αγορά και η εμπορική της πολιτική θα έχει να παίξει ένα αναμφισβήτητο ρόλο σχετικά. Ευχαριστώ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος, και θα, ξαναδώσω τώρα προηγουμένω το λόγο στην Κομισιόν, πρωτού πάω στην εισηγήτρια. Κυρία Ότμαϊερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αξιότιμα μέλη της Επιτροπής του Κοινοβουλίου για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα βοηθήσει πολύ τη, τη δουλειά μας στην υπηρεσία. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και την ευκαιρία να απαντήσω και να πάρω το λόγο. Συνολικά η Επιτροπή καλωσορίζει το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής σας. Έχετε θετική αξιολόγηση του σχεδίου Juncker, του επενδυτικού σχεδίου και κυρίως του εξωτερικού του σκέλος, σκέλους. Να σας δώσω κάποια στοιχεία για το που βρίσκεται μέσα σε ένα χρόνο κινητοποίηση 127,2 δις ευρώ για επενδύσεις σε διάφορα κράτη-μέλη. Θα υποφεληθούν 290.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Μπόρεσε το ΕΦΣΙ να προσελκύσει και άλλες πηγές επενδύσεων που είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Περίπου τα 2 τρίτα της συνολικής επένδυσης προέρχεται από τους ιδιώτες επενδυτές η πρόταση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Σεπτεμβρίου να παρατείνει και να επεκτείνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων μέχρι το τέλος της παρούσας προγραμματικής περίοδου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου συμπεριλαμβάνει αυτό, αυτή τη συμβουλευτική θερμοκοιτίδα για να έχουμε τεχνική βοήθεια και μάλιστα και δι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη γίνονται συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο για το πώς θα συμμετέχει κανείς στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, μιλώ για την, Κίνα, για την Κίνα, για τις τρίτες χώρες, η Κίνα ήταν η πρώτη που απλά εξέφρασε τη βούλησή της να συμμετάσχει. Ακούγοντας τη συζήτηση είναι σημαντικό να διευκρινίσει κανείς ότι το εξωτερικό σκέλος δεν είναι επέκταση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι ένα νέο σχέδιο που έρχεται ως συνέχεια του ΕΦΣΥ. Είναι προσαρμοσμένο στις ε, ανάγκες των γειτονικών χωρών και των αφρικανικών χωρών με πάντοτε γνώμονα την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και την επίλυση του μεταναστευτικού Θέλουμε να προσελκύσουμε τους ιδιώτες επενδυτές, τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να στηρίξουν έργα που δεν θα είχαν χρηματοδοτηθεί παλαιότερα. Και άρα ισχύει η αρχή της προστατικότητας. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω Κάπου εδώ να ολοκληρωθεί ο κατάλογος των επιπρόσθετων ταμείων. Μου δημιουργεί πρόβλημα, για να σας το πω με πάσα ειλικρίνεια, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργεί ταμεία για τα πάντα και άρα αυτά να είναι εκτός ελέγχου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ειδικότερα εάν αυτά τα ταμεία περιλαμβάνουν τμήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και αν αυτό ισχύει, δεν υπάρχει καμία δημοκρατική νομοποίηση για την ύπαρξη ε, των ταμείων αυτών. Επομένως, δεν είμαι φίλος ε, της πληθώρας, του πληθωρισμού ταμείων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε προς τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ένας από τους στρατηγικούς ε, στα, στόχους του ΕΦΣΥ είναι να προωθήσει την ε, απασχόληση και τη μεγέθυνση. Αλλά κάθε φορά που έρχεται ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν για να μας δώσει <clears throat> πληροφορίες για τα βασικά στοιχεία, ποτέ δεν μας λένε στοιχεία απασχόλησης. Θα ήθελα να ξέρω ποιο ήταν το αποτέλεσμα των σχεδίων όπω έχει συμμετάσχει το ΕΦΣΥ, πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί και πού. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι σημαντικά τα στοιχεία για τη δημιουργία της απασχόλησης, αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι όταν μιλάμε για σχέδια μεγάλων υποδομών που είναι 75% της λειτουργίας του ΕΦΣΥ, δεν βρισκόμαστε ακόμα στη φάση εφαρμογής. Όταν τα σχέδια αυτά πάρουν έγκριση για χρηματοδότηση, θα δούμε στα επερχόμενα χρόνια την αύξηση της απασχόλησης. Δεν μπορώ να σας δώσω λοιπόν στοιχεία για την απασχόληση αυτή τη στιγμή. Θα σας απασχολήσω. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργεί ένα υπόδειγμα, ένα μοντέλο για να αξιολογήσει την, ε, τον αντίκτυπο στην απασχόληση που μπορεί να σας δοθεί του χρόνου. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 5 η Οκτωβρίου για τον πρώτο χρόνο της, ε, του ΕΦΣΥ μπορεί να σας πληροφορήσει και θα υπάρξει και μια περαιτέρω αξιολόγηση η οποία θα συμβάλλει στην διαδικασία αξιολόγησης που ξεκίνησε από τις πρώτες προτάσεις της Κομισιόν στις 14 Οκτωβρίου. Αυτή η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα είναι έτοιμη στα μέσα Νοεμβρίου. Παρακαλώ. Νομίζω ότι η εκπρόσωπος της Κομισιόν, λέει κύριος Ντάτμουθ, είναι κάπως ταπεινόφρον σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το ταμείο αυτό δημιουργεί πολύ καλοπληρωμένες δουλειές για αυτούς που δουλεύουν για το Ταμείο Εύση. Πόσες θέσεις λοιπόν δημιουργήθηκαν για τους εργαζόμενους στο Ταμείο Εύση. Α, αυτοί όμως οι οποίοι δεν δουλεύουν στο Ταμείο δεν ξέρουμε καθόλου αν έχει δημιουργηθεί κάποια θέση επασχόληση. Αλλά αν μας πει η Επιτροπή πόσα άτομα δουλεύουν στο Ταμείο αυτό, πόσο πληρώνονται και πόσα παίρνουν μεικτά. Αν δεν έχετε αυτά τα στοιχεία θα σας έλεγα πρέπει να μας τα φέρετε κάποτε. Παρακαλώ. I would suggest, uh, Θα προτιμούσα να σας δώσω τα στοιχεία αυτά εγγράφως. Μα τι σημαίνει αυτό, λέω ο κύριος Ντάρτμουθ. Ε, δεν μου άρεσε η ερώτησή σας και δεν την απαντήσω. Τι ακριβώς σημαίνει η απάντηση που μου δώσατε. I'm my the chair. Uh, no, I don't, don't. Ρωτώ Το ταμείο αυτό το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μπορούν θα θαυμάσια να σας δώσουν στατιστικά στοιχεία για το πόσα άτομα συμμετέχουν στην ε, υλοποίηση αυτού του ταμείου θα ε, έπρεπε να το κάνουμε. Θα ζητήσω από την Κομισιόν να μας δώσει κάποια στοιχεία για το πόσα άτομα βρίσκονται ε, απασχολημένα στην ε, υλοποίηση του Ταμείου και ποιες είναι και οι αποδοχές τους. Ευχαριστώ. Εμμανουέλ. Ευχαριστώ. Δεν θα συμμετάσχω στη συζήτηση που ξεκίνησε ο κύριος Ντάρθμουθ. Βλέπω ότι φεύγεται ούτως ή άλλως. Άλλωστε το Μένο Βασίλειο φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επομένως δεν θα σας αφορά το θέμα λίαν συντόμως. Ή στο επανειδήν ή μάλλον αντίο. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι ο κύριος Ντάρθμουθ μόλις αποχώρησε από την αίθουσα θέλει το σκληρό Brexit. Να επανέλθω σε αυτό που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, γιατί θέσατε ένα πραγματικό ερώτημα. Θέλησα να το βάλω αυτό που είπατε μέσα στην έκθεση, αλλά είναι κάπως περίπλοκο. Ακούγοντας τους συναδέλφους, θεώρησα ότι είναι υπέρ τέτοιου, τέτοιων πρωτοβουλειών. Όμως η παρατήρησή σας αξίζει να σταθούμε λίγο περισσότερο, γιατί ε, ε γύρει διάφορα ερωτηματικά και συμφωνώ απολύτως. Τώρα, για τις εξωτερικές επενδύσεις, συμφωνώ με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι για τη μετανάστευση, για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Ευρώπης να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες ούτως ή άλλως για να ξεφύγουν από τη φτώχεια, για να επιλύσουν διάφορες διαρθρωτικές ε, δυσκολίες είναι υποχρέωση της Ευρώπης, δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη ε, ε, συζήτηση λόγω συγκυρίας. Είναι πάγια υποχρέωση της Ευρώπης αυτή. Επομένως δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Αντιθέτως πιστεύω ότι είναι πολιτικό εγχείρημα, πολιτική αποστολή της Ευρώπης να βοηθήσει δομικά ε, όλες αυτές τις χώρες με τις οποίες μας συνδέουν δεσμοί ε, φιλίας και οι οποίες αντιμετωπίζουν θεαματικές κρίσεις. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμφωνούμε όλοι για τη διάγνωση. Πρέπει να τις ενισχύσουμε για να γίνουν πιο διεθνείς, να τις βοηθήσουμε να εξάγουν περισσότερο, να στραφούν προς τον υπόλοιπο κόσμο. Είμαι έτοιμος να έχω συζήτηση μαζί σας, κυρία Κέλλερ. Ε, στρατηγική συζήτηση για το πώς πρέπει να τοποθετηθούμε, ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι μηχανισμοί βοήθειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ δεσμεύομαι να κάνω αυτό το διάλογο μαζί σας και με, πας, ε, με κάθε ενδιαφερόμενο. Για την Κίνα, να πω ότι δεν είναι ο στόχος μας να παρεμποδίσουμε την Κίνα να βάλει χρήματα, αλλά να ε, μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι Κινέζοι να μην έχουν προνόμια στη διακυβέρνηση και στη διαχείριση. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες σε επίπεδο Ευρώπης για την εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσο ό,τι αφορά την Κίνα και όσο ευρωβουλευτές είναι καθήκον μας να είναι οι πάντες ενήμεροι. Και δεν μιλάω μόνο για την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες θέλησαν να μπουν σε αυτό το ταμείο και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν το λέω για να στιγματίσουμε τη χύψη χώρα αλλά θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, επιβεβαιώσει ότι επαγρυπνά ε, για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους μισθωτούς και τους ε, καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Προθεσμία λοιπόν για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 17η Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 9 και 10 Νοεμβρίου. Το τελευταίο θέμα για σήμερα είναι το 11. Ετήσια έκθεση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χρηματοδοτική δράση. Ο κύριος Ζαντό δεν είναι παρόν που είναι ο εισηγητής. γιατί προετοιμάζει την υποψηφιότητά του ως Προέδρου της Γαλλίας εξ ονόματος των Πρασίνων. Ελπίζω να τα καταφέρει να είναι ο υποψήφιος των Πρασίνων. Καλή τύχη. Και η Σκά Κέλλαρ έχει το λόγο. Θα μεταφέρω τις καλύτερες ευχές σας στον κύριο Ζαντό. Ο Γιάννη λοιπόν μου ζήτησε βασικά να διαβάσω τη δήλωσή του θα προσπαθήσω να το κάνω. Λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη από τις συζητήσει σήμερα για την γνωμοδότησή μας για την ετήσια έκθεση 15 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εγώ θέλω να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία που είχαμε πέρυσι για την αντίστοιχη διατύπωση για το 14 κατά κάποιο τρόπο ίσως είναι δύσκολο να επαναληφθεί η επιτυχία της προηγούμενης προσπάθειας. Η γνωμοδότησή μας για το 2014 υπερψηφίστηκε με δύο αποχές και χωρίς μία ψήφο κατά. Και αυτό έδειξε την εκτίμησή μας στην εργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Περιλαμβάνει 25 λεπτομερείς συστάσεις που εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και για τη φετινή γνωμοδότηση. Η ενδιάμεση αναθεώρηση για τις δραστηριότητες της τράπεζας δεν είχε βέβαια ολοκληρωθεί και πάρα πολλές ε, ε, αναφορές σχετικά με την συνεργασία με το Στρατηγικό Ταμείο δεν είχαν δημοσιευθεί. Μέσω τροπολογιών όμως ε, θα υπάρξουν αρκετές τροπολογίες που θα ενημερώσουν το κείμενο και το ίδιο θα κάνω και εγώ με τις δικές μου. Να αναφερθώ λίγο στις προτάσεις τις οποίες κάνω. Στην παράγραφο 1 απλά σημειώνω πώς έχουν τα πράγματα. Αναφέρομαι στο ε, βασικό έγγραφο για το προσανατολισμό της τράπεζας αυτής, δηλαδή η εντολή την οποία θα δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εξωτερικό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα πρέπει να είναι συμβατός με τους στόχους αηφορίας για των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζω ότι θα υπάρξει δυνατότητα να διαβάσουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην παράγραφο 2 υιοθετούμε το βασικό αίτημα της προηγούμενης νομοδότησής μας ένα σύστημα δηλαδή που θα αναφέρεται στον σεβασμό της τράπεζας στις βασικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Ελπίζω ότι στο εσωτερικό αυτής της ενδιάμεσης αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα της βελτίωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών μάλλον ανάμεσα στην Τράπεζα και την Επιτροπή και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και για τη μετανάστευση. Η ενδιάμεση αξιολόγηση επίσης λέγει ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές της τράπεζας. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες ενδείξεις που θα μπορούμε εμείς να ελέγχουμε την συμβατότητα των αποφάσεων της τράπεζας με το άρθρο 21. Η παράγραφος 3 συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκινήσαμε τον προηγούμενο χρόνο έτσι ώστε να είναι ηγητική τράπεζα ή συγκεκριμένη στον δανεισμό προγραμμάτων για δράση στον τομέα του κλίματος. Έχει όμως τεράστιες επίσης ποσότητες χρηματοδότησης και στα ορυκτά καύσιμα και μετά από το COP21 θα πρέπει να σταματήσουμε ουσιαστικά να επιδοτούμε τα ορεικτά καύσιμα. Η παράγραφος 4 και αυτή διαπιστώνει το πώς έχει η κατάσταση και λέγει ότι θα πρέπει η δράση αυτή να βοηθήσει και να ενσωματωθεί και στο νέο Ταμείο για την Αφρική. Η χρηματοδότηση του νέου αυτού μέσου θα πρέπει να λάβει υπόψη και την αρχή της προσθετικότητας. Εδώ όμως θα πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο. Ελπίζω να το κάνετε και μέσω των τροπολογιών σας. Παράγραφος 5 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Λατινική Αμερική. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα έχει να παίξει ένα κεντρικό ρόλο για τη στήριξη των μικρομεσαίων, θα συμφωνήσουμε πλήρως εδώ, και η παράγραφος 6 θέτει ένα άλλο θέμα για το οποίο απαιτείται περισσότερη έρευνα και θα μας απασχολήσει και στην Επιτροπή μας τα επόμενα χρόνια. Συνεργασία δηλαδή ανάμεσα στην τράπεζα αυτή και τη νέα Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Θα θέλαμε ε, να συμμετέχει το Ταμείο αυτό και στα πλαίσια του καινούριου αυτού στρατηγικού ταμείου και θα πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε στο κεφάλαιο της επενδυτικής αυτής ασιατικής τράπεζας αλλά δημιουργούνται αρκετά πρακτικά θέματα ε, τα οποία έχουν σχέση με τον εντελώς διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης των δύο πιστοτικών οργάνων. Η AAIB ε, θα παίρνει αποφάσεις ε, που δεν θα επηρεάζονται ουσιαστικά από το Διοικητικό της Συμβούλιο, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Και δεν θα θέλαμε εμείς να χρηματοδοτούμε μια τράπεζα η οποία ενισχύει και επιδοτεί την πυρηνική ενέργεια ή την επεξεργασία προϊόντων άνθρακα, εξόριξης άνθρακα. Ελπίζω λοιπόν να συνεργαστείτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τροπολόγησης. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα στον, ε, ε Γιάννη και τώρα ο κύριος ε, Τσίκα είναι ο πρώτος, Τσίκου είναι ο πρώτος ο οποίος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση του κύριου Σαντό. Μου φαίνεται μια καλή πρόταση. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί του, ιδιαίτερα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, όπως ε, η ανάγκη που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να λειτουργεί με συμβατό τρόπο ε, με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την αηφορία και στην παράγραφο 4 να εμείνει στα θέματα της χρηματοδότησης προγραμμάτων για το κλίμα. Ε, θα πρέπει να δούμε όμως τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα της διεθνοποίησης των μικρομεσαίων. Είναι λίγες οι μικρομεσαίες ακόμα, οι οποίες έχουν την δυνατότητα χρηματοδότησης για την διεθνοποίηση της δραστηριότητάς τους προς τρίτες αγορές. Έχουμε τους ίδιους περιορισμούς για την πρόσβαση στην διεθνή αγορά, αν και αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο τον οποίο παίζει η συγκεκριμένη τράπεζα και, στις, και για τις επιχειρήσεις των 28 χωρών. Πρέπει λοιπόν να γίνουν περισσότερα. Πρόσβαση λοιπόν στην πίστοση, εκτός από το να υπογραμμίζει όπως έχουμε δει στο παρελθόν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο σκελετός της ευρωπαϊκής οικονομίας, να πούμε ότι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι ένα βασικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα έτσι ώστε οι μικρομεσαίες που δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν προγράμματα ανταγωνιστικά των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων να έχουν προτεραιότητα στην χρηματοδότηση από τους ενδιαμέσους χρηματοδοτικούς φορείς και να την χάνουν επίσης και συνδρομής για την σωστή αίτηση χρηματοδότησης. Αυτό θα βοηθήσει με δύο τρόπους. Πρώτον, θα οδηγεί στην χρηματοδότηση προγραμμάτων που θα γίνουν πλέον πραγματικότητα και δεύτερον θα εφαρμόζει και θα βελτιώνει την διαχείριση των επαφών ανάμεσα στην μικρή αυτή επιχείρηση και στις τοπικές πιστοτικές αρχές, οι οποίες θα συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα διοχετεύουν στην τοπική οικονομία την ρευστότητα την οποία έχει στη διάθεσή της η Τράπεζα η Ευρωπαϊκή. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της επικοινωνίας. Πάνω σε αυτό θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Εγώ προέρχομαι από κάποια εδάφη στα οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τοπικές τράπεζες ενδιαμέσους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δεν γνωρίζουν ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Υπάρχει μια στρέβλωση της πραγματικότητας. Υπάρχει μια ανησυχητική έλλειψη ενημέρωσης ε, και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει καθήκον εδώ σωστής ενημέρωσης. Εμείς ε, θα πρέπει ε, να δείξουμε ότι ναι μεν λειτουργούν με, με διαμέσους, αλλά υπάρχει δυνατότητα να ξεπεράσουν τις δυσκολίες επικοινωνίας. Λοιπόν, υπάρχει σκεπτικισμός και κριτική των μικρομεσαίων απέναντι στην Ευρώπη που επολύσαν φίλεται στην έλλειψη ενημέρωσης. Πολλές φορές οι ενδιάμεσοι υποχρεώνονται να στέλνουν μια επιστολή στις επιχειρήσεις ενημερώνοντάς τους ότι τα χρήματα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της διαφάνειας. Εμείς α, ε, ε, θεωρούμε θετικές τα ε, προτάσεις της ΜΕΗ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη βελτίωση της διαφάνειας και νομίζω ότι από τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιμείνουμε σε υψηλή ε, εταιρική ευθύνη έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση ε, για τον προϋπολογισμό και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Τώρα, για την ίδια τη δομή θα ήθελα στο κείμενο της γνωμοδότησης να προστεθεί μία παράγραφος για τις δραστηριότητες χρηματοδότησης των υποδομών. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στις ε, περιφέρειες της Ευρώπης. Εκεί υπάρχουν ε, πολλές φορές πολύ υψηλοί γεωγραφικοί περιορισμοί και χάρη σε υψηλής φιλοδοξίας χρηματοδοτήσεις μπορεί να επιτρέψουμε να βελτιωθούν οι εμπορικές συναλλαγές. Δηλαδή, Σικελία με την Αραβική Χερσόνησο ή με τη βόρεια ακτή της Αφρικής. Ροντρίγες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι καλώς εξετάζουμε τις δύο σχετικές εκθέσεις γιατί πρέπει να συντονίσουμε την θέση μας και για τα δύο θέματα. Συμφωνώ με τον κύριο Μορέλ απολύτως και συμφωνώ και με τον εισηγητή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πολύ σωστά παρουσιάζει τα στρατηγικά σημεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εμάς, το ότι τηρούνται οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, οι στόχοι αυτοί, να είμαστε πιο φιλόδοξοι στη νέα στρατηγική καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, να πω ότι συμφωνώ με τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ πρέπει να φτάσει η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μου μου λένε πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Είναι παντελής η απουσία ενημέρωσης για το ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι πολύ σημαντικό να γίνουν γνωστά όλα αυτά που γίνονται, ότι μπορούμε να διευκολύνουμε κεφάλαια για όσους έχουν επενδυτικά σχέδια και Εάν έχετε ε, και αν έχετε στοιχεία να τα μοιραστούμε, εγώ θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Ε, για παράδειγμα, για τη διαφάνεια. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς τους λόγους για τους οποίους απορρίπτεται το αίτημά του ε, για χρηματοδότηση. Να υπάρχει διαφάνεια και για τους λόγους για τους οποίους δόθηκε και για τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε. Γιατί αν δεν ξέρουμε ε, γιατί απορρίφθηκε ένα συγκεκριμένο έργο, τότε δύσκολα θα παρουσιάσουμε επόμενο έργο υποψήφιο. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν τις, αιτίες, τις αιτίες. Και πρέπει να κάνουμε περισσότερα στην ε, ε, απλούστευση, τοπικό χαρακτήρα, τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό να έχουμε υπόψη μας. Αυτές πρέπει να αναπτυχθούν και να επενδύσουν και για να μείνει ο κόσμος στις κοινότητες, στους δήμους. Επομένως η τεχνική βοήθεια είναι πολύ σημαντικό. Και τέλος, πολύ σημαντικό είναι τα κριτήρια επιλογής. Πώς θα διαλέξει κανείς ε, τα, τις επιχειρήσεις. Δεν αρκεί να υπάρχουν έργα που να σέβονται, να τηρούν ε, τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και το καθεξής. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυτές τις επενδύσεις πρέπει να διέπονται από εταιρική ε, κοινωνική ευθύνη και να έχουν δεσμευτεί γι' αυτό. Και να έχουν δεσμευτεί στη βασική αρχή για ίσο, ίση εργασία, ίσο μισθό. Δεν μπορούμε να έχουμε διακρίσεις. Και τέλος, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να απευθύνω ένα ερώτημα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων καταρχάς. Ναι, καλώς. Τότε θα ήθελα ε, και σε εσά να απευθύνω το εξής ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να υπάρχει μεγαλύτερη όθηση των επενδύσεων συμφωνήθηκε αυτά να μην μπουν στο έλλειμμα των χωρών. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τα επενδυτικά έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και που προωθούν οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις που έχουν ίδιους στόχους, δηλαδή να έχουν μεγαλύτερη επενδυτική διαφοροποίηση. Αυτά γιατί να μετρήσουν για το έλλειμμα και για το χρέος αφού πληρούν τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών έχει απορρίψει έργα ε, γιατί θα έπρεπε η επένδυση να συνυπολογιστεί για το έλλειμμα και το χρέος. Στην περιφέρειά μου αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Είναι ένα κριτήριο από το οποίο δεν μπορείτε να παρεκκλίνετε σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ζαντό, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο υποψήφιος των Πρασίνων στην ε, γαλλική προεκλογική εκλογή. Αυτό θα, να, θα αναμοχλεύσει λίγα τα πράγματα στη Γαλλία. Θα ανακατεύσει την τράπουλα. Για την έκθεση αυτή έχω απλώ μερικέ προτάσει που δεν πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενε. Είναι κάτι που απορρέει από την κοινή λογική για αυτά τα οποία θα μπορούσαν να προσθεθούν στην έκθεση αυτή. Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει περισσότερα για να εξασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει σαν στόχο αυτέ οι επιχειρήσει να μπορούν να ενταχθούν στην συνολική αλυσίδα προμήθειας και να αυξήσουν την κλίμακά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ιδίω στι χώρε που έχουν προτιμησιακά καθεστώτα εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να θα του δώσει λοιπόν μεγαλύτερε ευκαιρίε για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Δεύτερον, Χαιρετίσουμε την έκκληση του εισηγητή η δράση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνάδει με τι αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, <clears throat> μεταξύ αυτών τις αρχές μιας ανταγωνιστικής και τίμιας οικονομίας της αγοράς και το ελεύθερο εμπόριο. Πρέπει λοιπόν τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων να μην πηγαίνουν μοναχά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε λογικές ε, αναπτύξεις υποδομών και επομένω που μπορούν να δράσουν, γιατί χωρί αυτήν την υποδομή πολλά αναπτυσσόμενα κράτη δεν μπορούν να αναπτύξουν τα προϊόντα του και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν και να πολλούν αγαθά από και προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσω η γνωμοδότηση μπορεί να υπογραμμίσει αυτήν τη σύνδεση και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει περισσότερα σχετικά. Τρίτον, πιστεύω, ελπίζω, θέλω να συμφωνήσουμε όλοι για το θέμα αυτό, να τροποποιηθεί η γνωμοδότηση ώστε όλες οι δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να λάβουν υπόψη την ανάγκη να υπάρχει συνεχής και μόνιμη εμπλοκή των ενδιαφερομένων και το υψηλότερο επίπεδο ε, διαφάνειας, όπως είπε και η συνάδελφός μας από τους σοσιαλιστές, είναι απαραίτητο τα ταμεία αυτά, τα κονδύλια των κάποιων μελών, να διέπονται από το υψηλότερο επίπεδο λογοδοσίας και αποτελεσματικότος, Τέταρτο και τελευταίο, να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι ο μόνος μεγάλος δανειστής που είναι ενεργός εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συνεχίσει να δημιουργεί συνδέσμους με την Αφρικανική και Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης ώστε να βρουν συνέργειες, συνέργειες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε επιμερισμό πόρων και να εξασφαλίσουν ότι οι δραστηριότητε όλων αυτών των φορέων δεν είναι σε ανταγωνισμό αλλά συνεργατική. Και θέλω να ε, εκφράσω την ικανοποίησή μου για την παρουσία του εμπειρογνώμονα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Επενδύσεων και θέλω να το ρωτήσω αν υπάρχουν και ενδιαφέρουσε εξελίξει στον τομέα αυτό. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε τι δραστηριότητε αυτή τη στιγμή αναλαμβάνονται για να επιτευχθεί η συνεργασία με αναπτυξιακές τη Αφρική και τη Αμερική. Ο κύριο Τάκουλα για τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με... Μου δημιουργεί έκπληξη αυτό, αλλά λέμε στη Φιλανδία δεν θα προσθέσω πολλά γιατί δεν είμαι και ο σκιώδης εισηγητής αλλά ήμουν παρόν σε μια συζήτηση όπου αναφέρθηκε αυτή η ανησυχία σε σχέση με τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλο <clears throat> δυναμικό αν θέλουμε λοιπόν να οικοδομήσουμε την Ευρώπη με αηφόρο τρόπο δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο αλλά επειδή μου είπατε ε, μου δώσατε το λόγο. Θέλω να ευχηθώ στο Γιάννη κάθε επιτυχία στον αγώνα του για την εκλογή του στην ε, ε, Γαλλική Προεδρία και φαίνεται ότι είναι πολλοί που είναι αντίπαλοι του για, το, για τη θέση αυτή. Αυτά ήθελα λοιπόν να πω, να ευχηθώ και πάλι στο Γιάννη. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα το ουσιαστικό εκτός αυτών. Ευχαριστώ πολύ, και ο πρόεδρος, ο κύριος Τάκμουθ. Είναι κάπως ε, ταπεινόφρονο ο κύριος ε, Τάκουλα, αλλά αυτά που είπε είναι πολύ χρήσιμα. Μα δεν ξέρω αν είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσθέσουν αξία σε αυτή την έκθεση, ακόμα και εγώ ίδιος. Επαναλαμβάνω <clears throat> αυτά τα οποία είπαν και οι άλλοι. Εύχομαι στον κύριο Ζέντο κάθε επιτυχία στην προσπάθειά του να είναι ο υποψήφιος για τη Γαλλική Προεδρία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είχα την τιμή, αν μπορεί να θεωρηθεί τιμή, να γράψω μια παράλληλη γνωμοδότηση πριν από πολλά χρόνια και διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ακολουθεί γραμμές εμπορική τράπεζας σε πολύ μεγάλο βαθμό και ίσως μπορεί να με, μου τα επιβεβαιώσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ότι δεν έχει βέβαια επισφαλή δάνεια αλλά όσο περισσότερο τους ε, επιβάλλουμε μη εμπορικούς στόχους τόσο πιο πιθανό είναι ότι θα αυξηθεί το επίπεδο ή θα υπάρξει ένα επίπεδο επισφαλιών στην τράπεζα αυτή. Υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία θέλουμε να πετύχει τον Α και τον Β στόχο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα αλλά θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι πάντα με αδίδυτο τρόπο θα υπάρχει ένα κόστος σε κάποια σε όλες αυτές τις Δεν κατάλαβα πολύ καλά, δεν άκουγα τη μετάφραση. Το ε, Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα μερίδιο κατά 16,1 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 39 δισεκατομμύρια περίπου. Μέχρι ότου βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάμε πίσω τα λεφτά μας, που είναι κάποια χρόνια μπροστά, όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επίση, ό,τι αφορά την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να λειτουργήσει ω εργαλείο τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια πολιτική, και αυτό θα το αφήσω κατά μέρο, τότε πράγματι δεν τη επιτρέπει αυτό να λειτουργήσει ω μια επωφελή τράπεζα. Και το τρίτο σημείο, και θα σα τα λέω πάρα πολύ σύντομα, λέει το τρίτο σημείο, ζητά από την Κομισιόν να υπάρξει ένα φιλόδοξο ε, πρόγραμμα για την εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων. Μήπως είναι αυτό κάτι που πρέπει να κάνουν οι μηχανικοί του περιβάλλοντος και όχι αυτοί που είναι μπροστά από ένα υπολογιστή στο Λουξεμβούργο. Και το ίδιο ισχύει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο εκπρόσωπος της ομάδας του ΕΛΚ, ο σκιοδησίτης του ΕΛΚ, το είπε πολύ καλά. Όλοι υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την... πρέπει να Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Το πρόβλημα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλες τις εταιρείε είναι να μπορούν να βρουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Όλες αυτές οι σκέψεις είναι καλή ευσεβής πόθη, αλλά μπορούμε να έχουμε κάποιες στατιστικές για το ποσοστό και σε νούμερα και σε αξία δανείζονται στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην πίστοση. Δεν συμφωνούμε πολύ με τους πράσινους, αλλά συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει διαφάνεια. Και για τη διαφάνεια το θέμα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το ποσοστό των δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τέλος η Ασιατική Τράπεζα Υποδομών η Τράπεζα Επενδύσεων για τις υποδομές στην Ασία ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί από την Κίνα ως αντίβαρο στην Παγκόσμια Τράπεζα και ως ε, όχημα για να αυξηθεί η επιρροή της Κίνας στο οικονομικό χώρο. Και ο Λευκό είπε ότι μετά από πολλέ συζητήσει έχουμε εξετάσει κατά πόσον η Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών της Ασίας θα πετύχει τα υψηλά πρότυπα σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και επίπεδο διακυβέρνηση. Αντί λοιπόν να προχωρήσουμε αμέσως σε μια βεβαιασμένη συνεργασία με την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών, θα πρέπει να τεθούν ορισμένα ερωτήματα και τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να τεθούν στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει να τα θέσει και ο συντάκτης αυτής της νομοδότησης γιατί υπάρχουν σημαντικές ε, ανησυχίες για την Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών. Και τέλος, το τελευταίο τελικό μου σημείο είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα <coughs> Επενδύσεων έχει την έδρα στο Λουξεμβούργο που είναι η πλουσιότερη χώρα σε κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε, υπάρχουν 2.200 υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Λουξεμβούργο που θα ήταν καλύτερα να είναι σε μια πόλη όπως η, η Λιόν ή το Βουκουρέστι ή μια από τις πολλές πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα χαιρόταν να έχει 2.000 καλοπληρωμένους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου. Τώρα βλέπουμε ότι είναι 2.900 υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προσπαθώ να δω πόσοι από αυτού είναι πράγματι στο Λουξεμβούργο και ίσω ο τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μπορεί να μου το πει. Γιατί έχουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό φορέα, ο οποίος θα μπορούσε να πάει σε πολλές άλλες πόλεις της ε- Ευρωπαϊκή Ένωση. ακόμα και στην Λιψία. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πλουσιότερη, την πλουσιότατη με δίκτυο το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Θα πρέπει να συζητήσουμε σύντομα την, την έδρα των δύο ε, ευρωπαϊκών εξωτερικών υπηρεσιών που θα εγκαταλείψουν το Λονδίνο. Δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά δεν πρέπει να τα στείλετε στο Λουξεμβούργο. Ο κ. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ίσως μετά και στον εκπρόσωπο της Τράπεζας. Yes, from the Commission side, there are no additional... Δεν έχουμε κάποιο σχόλιο να κάνουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι ο συνάδελφος εδώ ίσως να θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Εγώ είμαι από την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ. Θα θέλαμε εμείς ε, να πούμε ότι συμφωνούμε με τις προτάσεις οι οποίες έγιναν για την έκθεση και για τις εξωτερικές δραστηριότητες Συμφωνούμε επίσης και με τους στόχους για την αηφόρο ανάπτυξη. Για τις εκθέσεις και αναφορές δεν μπορούμε να επιβάλλουμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται. Αλλά ό,τι κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα πρέπει να είναι συμβατό με τις αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής. Και βλέπουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί το άρθρο 19 για τον συνδυασμό των πόρων που χρησιμοποιούνται. Εμείς ε, συνδυάζουμε τις προσπάθειές μας σε διάφορες επενδυτικές προσπάθειες και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ό,τι γίνεται στον εξωτερικό τομέα να είναι συμβατό με τις εσωτερικές μας διαδικασίες. Υπήρξαν επίσης ε, συζητήσεις και για την βοήθεια προς τους μικρομεσαίες και νομίζω ότι είναι καλό να στρέψουμε το βλέμμα μας προς άλλες περιοχές του κόσμου. Επίσης ακόμα και θέματα μικροχρηματοδότησης μπορεί να καλυφθούν εν μέρει από την τράπεζα. Θα τα υποστηρίξουμε όλα σε αυτές τις προτάσεις. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν έχει να κάνει κάποιο σχόλιο. Ευχαριστούμε. Ίσως να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Εργάζομαι στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στις Βρυξέλλες. Όπως γνωρίζετε, μιλάμε για τον τρίτο πυλώνα, ο οποίος έχει σαν στόχο την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Οι κανόνες τους οποίους χρησιμοποιούμε πολλές φορές ε, όταν έχουν ελλείμματα σαν παράδειγμα μπορεί να μην δίνουν πρόσβαση στις μικρομεσαίες χρηματοδότηση. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και να αλλάξουμε κάποιους κανόνες. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς δεν πηγαίνει καλά σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχάς μέσω του διακανονιστικού πλαισίου το επενδυτικό περιβάλλον. Αυτό μπορούμε να κάνουμε από δικής μας πλευρά. Για τις μικρομεσαίες λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το θέμα για σας. Πόσες έχουν ενισχυθεί από πλευράς μας. Το 30% των δανείων τα τελευταία 2-3 χρόνια πηγαίνει στις μικρομεσαίες. Φτάσαμε σε 250.000 μικρομεσαίες το 2015. Πολλές από αυτές έχουν, οι περισσότερες από αυτές είναι μικροεπιχειρήσεις με κάτω από 10 υπαλλήλους. Σχετικά με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι μια πιστοτική, ένας πιστοτικός οργανισμός αν υπάρχει διαμεσολάβηση και άλλου πιστοτικού ιδρύματος υπάρχει πρώτα μια αξιολόγηση. Είναι δύσκολο βέβαια να πιέσουμε μερικές φορές ε, τις ε, τοπικές πιστοτικές δραστηριότητες να αναλάβουν κινδύνους σε χώρες όπως ε, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία όπου υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία για πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υπάρχει διαμοιρασμός κινδύνου με τα τοπικά πιστοτικά ιδρύματα. Για την έδρα της τράπεζας είπαμε ότι είναι στην Λουξεμβούργο Κοιτάξτε, αν ρωτήσετε τους συναδέλφους στο Λουξεμβούργο αν θέλουν να πάνε στη ή θα ενθουσιαστούν. Αλλά υπάρχουν θέματα στις συνθήκες τα οποία αποφασίζουν με διαφορετικό τρόπο. Και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω στη συνέχεια λεπτομερέστερες πληροφορίες. Και το αλικάντε καλό είναι λέει ο πρόεδρος. Υπάρχει μια επιπλέον ερώτηση. Ναι. Ε, μου απαντήσατε και θα ήθελα να μου πείτε εάν γνωρίζετε τις αιτίε για τις οποίες τα χρηματοπιστατικά ιδρύματα λένε όχι σε επενδυτικά έργα. Είναι λογικό να εμπιστευτεί κανείς τους αξιολογητές κινδύνου, τους αναλυτές κινδύνου, αλλά οι ίδιοι είναι που χρηματοδότησαν τη φούσκα. Μήπως είναι οι ίδιοι αυτοί που δεν διευκολύνουν επενδυτικά έργα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της φούσκας του κτηματομεσητικού κλάδου της οικονομίας, ε, δεν αποστρέφονταν καθόλου το κίνδυνο, ενώ τώρα τον αποστρέφονται πάρα πολύ. Και αυτό είναι περίεργο. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία δημοσίου τομέα και, εν πάση περιπτώσει, ισχύουν όλα αυτά στην περιφέρειά μου και δεν είναι και η μόνη και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να τα γνωρίζει και να έχει συμπράξει συνεργασίες δημοσίου ιδιωτικού ε, τομέα ε, για τα επενδυτικά έργα και να μην συνυπολογίζονται αυτά στο έλλειμμα και άρα ούτε και στο χρέο Θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ασκείται εποπτικά της καθήκοντα, όχι μόνο στο τι δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρυμάτα, αλλά και στο τι δεν δίνουν και γιατί είναι σε θέση να κάνει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει την τροποποίηση του νομοθετικού πλησιασίου, εάν αυτό τελικά περιορίζει τις δυνατότητες επιτυχίας των δράσεων αυτού του Ταμείου. Έχετε σχόλια, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι είναι μια ερώτηση επί της αρχής για το ε, χρηματοδοτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να πω ότι ούτε και εμένα με ικανοποιεί γιατί οι οικονομικοί περιορισμοί δεν είναι μοχλός για τη δημιουργία επενδύσεων και οι επενδύσεις είναι απαραίτητες στην περιφέρεια. Αυτό ισχύει και θα πρέπει αυτό να το απεικονίσουμε στη δράση μας, ειδικότερα ως, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η νεολαία είναι αρκετά ε, σκεπτική σε σχέση με την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης μεταξύ άλλων. Αυτό ήταν και το σχόλιο της ημέρας από ε, τη θέση του Προέδρου. Υπάρχουν παρατηρήσεις από τη σκιώδη συγγήτρια, την αναπληρώτρια συγγήτρια, κυρία Κέλλερ. Όχι. Θα μεταφέρουμε ε, στο Γιάννη όλα σας τα σχόλια. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, καταληκτική προθεσμία τροπολογιών 17 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και θα εξετάσουμε το κείμενο στη συνεδρίαση 9 και 10 Νοεμβρίου. Ε, θα εξετάσουμε τότε τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ όλους. Θα έχουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα και στις 6.30 θα ξεκινήσουν με ευθύ αμέσω με τον τριμερή διάλογο για τα όρυκτα από περιοχές συγκρούσεων.